I και κύριοι, καλή σας μέρα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους εγκαρδιότητα στη συνεδρίαση της ΣΥΤΡΕ. Έχετε λάβει την ημερήσια διάταξη, υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι. Δεν έχω ούτε ανακοινώσεις, οπότε μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στο σημείο 3 Τη ημερήσιας διάταξη τον εκτελεστικό οργανισμό για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και συζήτηση σχετικά με το σημερινό στάδιο του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, ΣΥΠ. Εκτελεστικός διευθυντής είναι ο κύριος Πατρίκ Λάμπερτ και έχουμε από, την, ε, ε, από τον οργανισμό αυτό τον Βίλιαμ Ζιλμπέρτ, την Πατρίς Γιόρντι και τον Χουσέιν Σατάφ. Ελπίζω να πρόφερα σωστά τα ονόματά σας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να καλωσορίσω φυσικά και τους συναδέλφους ε, που είναι παρόντες σε αυτή τη συζήτηση, την οποία θα πρέπει να ολοκληρώσουμε λίγο πριν τις 10, γιατί μετά έχουμε ψηφοφορίες. Κύριε Λάμπερτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμη ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε σήμερα τον εκτελεστικό μας οργανισμό και τα προγράμματά του. Γνωρίζω αρκετού ευρωβουλευτέ, αλλά είναι η πρώτη ευκαιρία που μα δίνεται να κάνουμε τέτοια επίσημα παρουσίαση στην Επιτροπή σα. Εγώ θα παρουσιάσω το σύνολο του οργανισμού μα και μετά οι συνάδελφοι θα σα δώσω κάποιε λεπτομέρειε για τα πιο ενδιαφέροντα για σας φαντάζομαι, προγράμματά, της. προγράμματά του. Συγγνώμη. Α ξεκινήσουμε με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική το 2020 έχουμε τις εμβληματικές πρωτοβουλίες στη διαφάνεια. Φαντάζομαι θα γνωρίζετε αυτές τις εμβληματικές πρωτοβουλίες, αλλά σας δείχνουμε τη διαφάνεια για να δείτε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο οργανισμός και τα προγράμματά του και πώς εμπλέκεται σε μεγάλο αριθμό αυτών των εμβληματικών πρωτοβουλιών. Θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για τον οργανισμό μας και το ρόλο του σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαράζει τις πολιτικές, είναι το σώμα που προσδιορίζει το πρόγραμμα εργασιών για τα προγράμματα και ο οργανισμός διαχειρίζεται τα διάφορα προγράμματα. Σημαντικό ζήτημα είναι ο διαχωρισμός μεταξύ του προγραμματισμού, των πολιτικών και της ε, εκτέλεσης. Αυτός ο διαχωρισμός είναι χρήσιμος και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την ε, και για τον οργανισμό που μπορεί να επικεντρώνεται στα βασικά καθήκοντα. Και μάλιστα το θέμα των πολιτικών, της χάραξης πολιτικών είναι σημαντικό σημείο της διαδικασίας. Σε ό,τι αφορά το χαρτοφυλάκιο του οργανισμού, βλέπετε στη διαφάνεια αυτή τα διάφορα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες, το Μάρκο Πόλο, την Ευρώπη για την Εφή Ενέργεια, την Οικολογική Καινοτομία και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τις, ε, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων. Οι συνάδελφοι σας αναφέρουν περισσότερα στοιχεία για το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, το ΣΥΠ. Γιατί εγώ θα επικεντρωθώ στα πιο γενικά στοιχεία για τον οργανισμό. Βλέπετε εδώ ότι έχουμε τα ίδια προγράμματα κάτω-κάτω στη διαφάνεια και βλέπετε και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς και τα σχέδια διαχειριζόμαστε, τα διάφορα projects. Αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε περίπου 550 projects στα διάφορα προγράμματα και ταυτόχρονα ε, στηρίζουμε περίπου 600 εταίρους στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων. Και μάλιστα κατά το τέλος των δημοσιονομικών προοπτικών θα έχουμε διαχειριστεί περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο όνομα φυσικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία παρόμοια και πάλι διαφάνεια. Εδώ έχουμε τα θέματα της ενημέρωσης της αναφοράς που πραγματοποιούμε προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε εκτελεστικός οργανισμός και διαχειριζόμαστε τα προγράμματα στο όνομα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κυρίως για συγκεκριμένες γενικές διευθύνσεις που είναι συγγενείς ε, όπως τις λέμε γιατί τη ε, Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Ω εκτελεστικό οργανισμό είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που αυτέ οι τέσσερι γενικέ διευθύνσει εμπιστεύτηκαν τη διαχείριση των προγραμμάτων του σε εμά, τον εκτελεστικό οργανισμό καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι τώρα, οι αποδέκτε αυτών των προγραμμάτων. Έχουμε ένα ευρύ μείγμα τέτοιων δικαιούχων Δικαιούχοι μπορεί να είναι επιχειρήσεις, οργανώσεις ε, επιχειρήσεων, δημόσιες αρχές, κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, όμιλοι, σωματεία, ενώσεις και ούτω Αυτό που θα ήθελα να τονίσω όμως είναι η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διαδικασία αυτή των προγράμματων των προγραμμάτων. Αν εξετάσουμε την πρωτοβουλία για την οικολογική καινοτομία, περίπου 65% των δικαιούχων αυτή τη οικολογική καινοτομία είναι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εφή Ενέργεια έχει αποδέκτε κατά 40% μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και σε ό,τι αφορά το ε, δίκτυο, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων, αυτό κυρίως ε, έχει ως ρόλο το, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δύο λόγια για την οργάνωση. Ε, εκτελεσ... Ε, κλασική οργάνωση με επιχειρησιακές δομές και δύο οριζόντιες δομές. Με τη διαφάνεια αυτή σας δείχνω την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα του οργανισμού. Όταν ξεκινήσαμε είχαμε μόνο ένα πρόγραμμα, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ζήτησε να διαχειριστούμε τρία επιπλέον προγράμματα, καταφέραμε να προσαρμόσουμε τη δομή μας πολύ εύκολα και ομαλά και πολύ υπεύθυνα ώστε να δημιουργήσουμε νέες μονάδες και να ανταπεξέλθουμε στις νέες μας ευθύνες. Άλλο σημαντικό σημείο είναι οι συνέργειες που ανέπτυξε ο οργανισμός μας μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων. Και έχω την αίσθηση ότι αυτές οι συνέργειες θα έμεναν ανεκμετάλλευτες αν τα προγράμματα αυτά εξακολουθούσαν να τα διαχειρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων το χρησιμοποιούμε για να προωθήσουμε και τα άλλα προγράμματα που διαχειριζόμαστε. Δηλαδή, φτάνουμε στις, στους αποδέκτες μας, α, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με αυτόν τον τρόπο μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων. Προσλάβαμε ένα μεγάλο αριθμό ειδικευμένου προσωπικού και εμπειρογνωμόνων και σήμερα έχουμε σχεδόν 150 υπαλλήλου, κυρίω συμβασιούχου, 80% είναι οι συνταξιούχοι και 20% προσωρινοί ε, υπάλληλοι με ε, συμβάσει περιορισμένου χρόνου και έτσι έχουμε καλύτερες σχέσεις και διασυνδέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε εμπειρογνώμονες σε στήριξη επιχειρήσεων, ενέργεια, περιβάλλον, μεταφορές, επικοινωνίες και ούτω καθεξής. Πρόσφατα μάλιστα κάναμε και μια αξιολόγηση του εκτελεστικού οργανισμού και θα ήθελα να σας αναφέρω μερικά πορίσματα αυτής της αξιολόγησης. Ε, ήταν ανεξάρτητοι οι εμπειρογνώμονες που ασχολήθηκαν με το έργο του οργανισμού και θεώρησαν ότι το μοντέλο της εξωτερικής ανάθεσης ήταν πολύ επιτυχημένο. Επίσης, οι πυρογνώμονε ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η διαχείριση των προγραμμάτων από τον οργανισμό ήταν αποδοτική και αποτελεσματική και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο οργανισμός αυτός παρέχει πολύ καλύτερο περιβάλλον ε, για την εφαρμογή του προγράμματος και έχει στενές επαφές με τους ε, δικαιούχους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα και το feedback που είχαμε από δικαιούχους και συμβαλόμενους ήταν πολύ θετικό μεγάλος βαθμός ικανοποίησης και από αυτούς. Ε, είχαμε 90 μέρες προθεσμία για την ε, καταβολή των ε, δόσεων των προγραμμάτων. Πολύ χρήσιμο αυτό και ιδιαίτερα χρήσιμο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνεχώς προσπαθούμε να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες. Και αυτό είναι σημαντικό για να μειώσουμε το διοικητικό άχθος για τους πελάτες μας που είναι κατεξοχήν μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως σας είπα. Βλέπετε στο οργανόγραμμα ότι έχουμε μια ειδική ομάδα, ε, μια ειδική μονάδα, συγγνώμη, που ασχολείται με την επικοινωνία. Αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τις ε, επικοινωνιακές μας προσπάθειες και μάλιστα αυτή η διαφάνεια συνοψίζει το έργο μας σε θέματα επικοινωνίας. Θα ήθελα να σας επισημάνω δύο-τρία σημεία. Τελευταία τριετία είχαμε περίπου 1 εκατομμύριο επισκέπτες στις ιστοσελίδες μας και μοιράσαμε περίπου 600.000 φυλάδια κατέτηση. Είχαμε 70, 700 συγγνώμη, κλιπ και 40 περίπου βίντεο τα επισκέφθηκαν 64 εκατομμύρια θεατές. Κάνουμε προσπάθειες να προβάλλουμε τα προγραμματά μας και κυρίως τα αποτελέσματά τους. Επίσης, ε, διαχειριστήκαμε και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας που έχει γίνει σημαντικό ραντεβού ετήσιο και τον Απρίλιο είχαμε 772 ε, ε, εκδηλώσεις σε 40 χώρες και πολλές συναυλίες και εκδηλώσεις έγιναν και στις Βρυξέλλες. Οπότε μπορούμε να συνοψίσουμε το έργο της, του εκτελεστικού οργανισμού λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν από εμά ένα υψηλό επίπεδο προδιαγραφών, ε, μια σωστή διαχείριση των προγραμμάτων, σωστή σχέση κόστους-οφέλους, μεγάλη προσαρμοστικότητα για να ανταποκριθούμε στις νέες συνθήκες και μάλιστα οι δικαιούχοι είναι ικανοποιημένοι γιατί λαμβάνουμε υπόψη ανάγκες τους και ε, προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε με ταχύ ρυθμό. Ένα άλλο συμπέρασμα από την αξιολόγηση των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Δεδομένης της ε, επιτυχούς διαχείρισης ε, και διεκπαιρέωση των προγραμμάτων από τον οργανισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτεται να αναθέσει και νέα προγράμματα στον οργανισμό μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μόλις πρόσφατα, χθε το απόγευμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε και την πρόταση για το μελλοντικό προπολογισμό. Οπότε το επόμενο στάδιο θα είναι ε, να διαχειριστούμε και να εκτελέσουμε σωστά αυτό το προπολογισμό. Και η τελευταία διαφάνεια ατενίζει το μέλλον. Ως οργανισμός θα συνεχίσουμε να θέτουμε την, τον οργανισμό μας στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών οργάνων και φυσικά στους πελάτες, ε, στους συμβαλόμενους και θέλουμε να υποστηρίξουμε τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής του 2020. Θα στηρίξουμε τα τρέχοντα και τα μελλοντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις ε, ε, περιβαλλοντικές κλιματικές πολιτικές, τις πράσινες τεχνολογίες και την καινοτομία. Αυτή είναι η ουσία και το έργο του εκτελεστικού μας οργανισμού. Θα δώσω τώρα το λόγο στου συναδέλφους που θα σα δώσουν περισσότερες λεπτομέρειε για τα επιμέρους προγράμματα, ξεκινώντας από τον Bill Gillard και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευθύνη Ενέργεια. So good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο συνάδελφος και εγώ είμαστε υπεύθυνοι για 500 τέτοια προγράμματα στον τομέα της ενέργειας, μεταξύ των οποίων και 18, τη δημιουργία 18 τοπικών υπηρεσιών ενέργειας. Ασχολούμεθα με την αποτελεσματικότητα στην ενέργεια, με την ενέργεια στις μεταφορές και με τις ανανεώσιμες πηγές και ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν και τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Εργαστήκαμε στην Επιτροπή πριν περάσουμε σε αυτή την υπηρεσία και νομίζω ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε καλύτερα στο εσωτερικό της υπηρεσίας αυτής από ό,τι λειτουργούσαμε στο Ευρωπαϊκό της Επιτροπής. Είναι ένα μη τεχνολογικό πρόγραμμα αυτό που έχουμε μπροστά μας για την ενέργεια, υποστηρίζει πολλές πρωτοβουλίες, οργανώνει και την εβδομάδα εν πάση περιπτώσει της βιώσιμης ενέργειας, τη συνάντηση των δημάρχων. Έχουμε ξεκινήσει πρωτοβουλίες οι οποίες είναι σαφέστατα κατανοητές στόχος αυτής της πολιτικής είναι να μετατρέψουμε την ομοθεσία και την πολιτική σε συγκεκριμένες δράσεις. Η πολιτική και οι οδηγίες μας καθοδηγούν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι επιχειρήσεις και οι πολίτες γνωρίζουν πώς να τις εφαρμόζουν. Γι' αυτό τα προγράμματα αυτά έχουν σαν στόχο να πετύχουν την καλύτερη κατανόηση του τρόπου εφαρμογής των κοινοτικών πολιτικών. Ποιε είναι οι βέλτιστες πρακτικές, τι είναι λειτουργικό και τι όχι. Υποστηρίζουμε ομάδες οργανώσεων στο εσωτερικό της Ένωσης που αυτό το στόχο έχουν και έχουν και τα κίνητρα για να τον επιδιώξουν. Παρέχουμε πληροφορίες, πληροφορίες της αγοράς και feedback σε αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις. Το πρόγραμμα ΙΗ έχει ένα προϋπολογισμό 730 εκατομμυρίων ευρώ για 7 χρόνια αυτό σημαίνει γύρω στα 100 εκατομμύρια κατέτος. Από το 2007 ο ετήσιος αυτός προϋπολογισμός αυξάνεται, αλλά οι δαπάνες για τα προγράμματα παραμένουν σταθερές. Αυτό σημαίνει, γίνεται γιατί από το 2009 τα χρήματά μας έχουν περάσει και από την Τράπεζα Ευρωπαϊκών Επενδύσεων για τεχνική βοήθεια προς δημόσιες αρχές στα πλαίσια των προγραμμάτων βιώσιμης ενέργειας. Υπάρχουν περίπου 3.000 εποφελούμενοι από τα προγράμματά μας σε 31, σε 31 χώρες. Οι περισσότερες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πάνω του 40%. Ένα χαρακτηριστικό πρόγραμμα είναι ένα με 2 εκατομμύρια για 2-3 χρόνια και εμπλέκει 8-9 οργανώσεις από διαφορετικές χώρες και υποστηρίζουμε μέχρι το επίπεδο του 75% δεν υποστηρίζουμε έρευνα και ανάπτυξη και τα χρήματά μας δεν χρησιμοποιούνται επίσης για την αγορά μηχανισμού, εξοπλισμών μηχανικών. Εμείς έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο το οποίο διαχειριζόμαστε και θα ακούσετε και από τη συνάδελφο περισσότερα σε λίγο. Τα προγράμματα της ΑΕΗ συμπληρώνουν τα ερευνητικά προγράμματα. Θέλουμε να επιταχύνουμε εμείς την ενσωμάτωση των αποδεδειγμένα χρήσιμων τεχνολογιών, λύσεων και πρακτικών. Να σας δώσω τρία παραδείγματα. Θέλουμε να μειώσουμε την γραφειοκρατία. Αν διαβάσετε την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές, λέει ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε οι διαδικασίες οι διοικητικές να γίνουν streamlined σε εθνικό επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό. Τι πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο, τι πρέπει να γίνει σε περιφερειακό επίπεδο, τι πρέπει να γίνει σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν ας πούμε προγράμματα για την αιωλική ενέργεια. Συμμετέχει η κυβέρνηση της Σκοτίας συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές και θέλουν ακριβώς μέσα σε ένα πρόγραμμα τριών ετών να μειώσουν κατά πολύ τη γραφειοκρατία. Ένα άλλο πρόγραμμα είναι το SF Energy Invest. Αυτό χρησιμοποιείται για την προώθηση των διαφορετικών ταμείων. Τα διαφορετικά ταμεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την βιώσιμη ενέργεια, αλλά οι στόχοι χρηματοδότησης δεν καλύπτονται. Εδώ έχουμε σαν ηγέτιδα θα έλεγα και συντονίστρια την Υπηρεσία Ενέργειας της Ολλανδίας και εκπροσώπους εννέα χωρών. Οργανώνονται συναντήσεις σε διαφορετικές χώρες εντοπίζοντας προγράμματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα διαφορετικά ταμεία. Συνάδελφοι της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακών Υποθέσεων συνεργάζονται μαζί μας. Το τελευταίο παράδειγμα είναι το EUREM για την βελτίωση των ικατοτήτων των διαχειριστών ενέργειας. Εφόσον είναι σωστά εκπαιδευμένοι καθιστούν τη βιομηχανία πιο ανταγωνιστική. Υπάρχει λοιπόν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τη Γερμανία το οποίο αντεγράφει θα έλεγα και σε άλλες 9 χώρες και κόστισε 24 εκατομμύρια. Συνεχίζεται μάλιστα το πρόγραμμα αυτό χωρίς τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άνω των 2.000 διαχειριστών στον τομέα της ενέργειας έχουν χρησιμοποιηθεί. Θα ήθελα να κλείσω με δύο επίσης καλά νέα θα έλεγα. Πρώτον, να πω ότι τα προγράμματα IEE e είναι δημοφιλή Έχουμε πάρει πάνω από 350 προτάσεις, μπορούμε να υποστηρίξουμε μόνο 50 ή 60, μία στις 6 δηλαδή. Και ένα άλλο καλό νέο είναι ότι ο έλεγχος αυτών οι οποίοι χρησιμοποιούν τα πλεονεκτήματά μας έδειξε ότι η διαχείριση των προγραμμάτων από τις ομάδες μας είναι κάτι το οποίο θεωρείται γενικότερα θετικό θα σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς τα προγράμματά μας βοηθούν να προωθηθούν οι πολιτικές στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας και της ανταγωνιστικότητας της ενέργειας. Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υποστηριχθούν οι ενεργειακές πολιτικές στα επερχόμενα δημοσιονομικά πλαίσια. Καλημέρα σας. Εγώ θα προσπαθήσω να σας δώσω μία μικρή γεύση από την οικολογική καινοτομία και το έργο της, του οργανισμού μας. Καταρχήν ο ορισμός. Έχουμε ε, επίτηδες ε, ευρύ ορισμό. Δεν περιλαμβάνει μόνο τις οικολογικέ επιχειρήσεις. Θα μπορούσε να είναι και ένας υποδηματοποιό ταγκάρι, οποιαδήποτε μικρομεσαία επιχείρηση που θέλει να αποκτήσει περισσότερο περιβαλλοντικό προσανατολισμό, να γίνει πιο πράσινη και να θέσει μια νέα υπηρεσία ή ένα αγαθό στην αγορά, εμπίπτει στον ορισμό. Δεν έχουμε μόνο τι οικολογικέ επιχειρήσει. Επίση έχουμε δύο πυλώνες ένα πυλώνα είναι επιχειρήσει και ο δεύτερο το περιβάλλον. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση όπω ξέρετε. Εμεί προσπαθούμε τι καλέ ιδέε να τι θέσουμε στην αγορά. Κάτι που είναι καλό και για τι επιχειρήσει, να είναι καλό και για το περιβάλλον. Τώρα πώ λειτουργεί αυτό το εργαλείο. Έχουμε το πρόγραμμα REACH που δεν είναι στόχος, δεν είναι υποχρέωση, δεν συνιστά νομική δέσμευση, αλλά έχουμε καταφέρει το 65% των δικαιούχων μας να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πολύ καλό στοιχείο αυτό για την υγεία και είναι σημαντικό μια υπηρεσία, ένα οργανισμό να έχει τόσο μεγάλο αριθμό δικαιούχων μικρομεσαίες επιχειρήσει. Και ακόμη πιο σημαντικό, 8 από τι 10 μικρομεσαίε είναι μικρέ και μικροσκοπικέ επιχειρήσει. Και έρχονται και προτείνουν ιδέες στην Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το κλειδί της επιτυχίας είναι η απλούστευση των εργαλείων και των μηχανισμών και επίσης μια σωστή ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που ενδιαφέρουν τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και η προσέγγιση είναι σημαντική. Δεν έχουμε αποκλειστικές προτεραιότητες. Οποιαδήποτε ε, φιλοπεριβαλλοντική ιδέα με δυναμικό αγοράς είναι σημαντικό. Ε, δεν έχουμε μεσάζοντες και αυτό είναι σημαντικό. Άμεση χρηματοδότηση μπορούν να έρχονται και να χτυπούν την πόρτα μας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει ελαστικότητα σε πολλές πτυχές. Φυσικά απαιτείται προστιθέμενη αξία για να, για να κατακυρωθεί ένα πρόγραμμα, αλλά δεν χρειάζεται να έχουμε και μια πολυεθνική εταιρεία ή όμιλο απέναντί μας. Και αυτό είναι σημαντικό για να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, έχουμε, λαμβάνουμε υπόψη ολόκληρο τον κύκλο της ζωής. Θέλουμε να είμαστε καλοί υδραυλικοί, να μην διορθώνουμε το σωλήνα σε μία πλευρά και να έχουμε διαρροή από την άλλη πλευρά λαμβάνουμε υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής, σημαντικό αυτό. Ούτε ζητούμε διοικητική άκαμπτη προσέγγιση. Θέλουμε να μας λένε οι επιχειρήσεις, ε, να μας διαβεβαιώνουν ότι έχουν λάβει υπόψη ένα συνολικό περιβαλλοντικό κριτήριο. Τώρα, τι γίνεται μετά την έρευνα και πριν την ε, θέση εμπορία της αγοράς. Χωρίς να έχουμε μια γραμμική προσέγγιση της καινοτομίας, είναι σημαντικό οι ιδέες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε επίπεδο πρωτοτύπου και επίδειξης να φτάνουν στην αγορά και μάλιστα 20% των προγραμμάτων προέρχονται από το, 7 από το 6ο ή 7ο ερευνητικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή από την Εθνική Έρευνα, το 20%. Τα υπόλοιπα από copyright, από ιδέες στην αγορά, από οποιαδήποτε πηγή. Έχουμε μία αιμονή με τη μόχλευση και την αντιγραφή από την αγορά. Θέλουμε έχουμε, να έχουμε ε, αποτελεσματική χρηματοδότηση, να υπάρχει μια συνέχιση, να αντιγράφονται ιδέες, να είναι αποτελεσματική η πόρη και φυσικά να πολλαπλασιάσουμε τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Ζητούμε από του δικαιούχου να βάζουν τι ε, ιδέε του στην αγορά. Αν δεν υπάρχει τέτοιο δυναμικό, δεν χρηματοδοτούμε προτάσει. Τώρα, με τι ασχολούμαστε. Το θέμα της αποτελεσματικότητας των πόρων είναι εγκάρσιο και πολύ σημαντικό. ανακύκλωση, πράσινες επιχειρήσεις, ε, τρόφιμα και ποτά, νερό, δομικά υλικά. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε. Υπάρχουν κάποιε γενικέ προτεραιότητε, αλλά δεν είναι εξαντλητικέ ή αποκλειστικέ έχουμε διάφορους τομείς, χεραμικά, κλωστεφαντουργικά. Δεν περιοριζόμαστε όμως σε συγκεκριμένους τομείς, απλώς έρχονται τέτοιες επιχειρήσεις και μας προβάλλουν τις ιδέες τους. Και έχουμε αρκετή επιτυχία στις εφαρμογές αυτές. Βέβαια υπάρχει και ένα τίμημα σε ό,τι αφορά ε, τη, τα ποσοστά απόρριψης, αλλά υπάρχει απορρόφηση των νέων καινοτόμων ιδεών στην αγορά. Όταν υπάρχει ανταγωνιστικό δυναμικό, υπάρχει απορρόφηση από την αγορά. Λοιπόν, και θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι ένα νέ, μια νέα φιάλη γάλακτος από ανακυκλωμένο χαρτί με ένα λεπτό πλαστικό, με μια λεπτή πλαστική επένδυξη, επένδυση, μικρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Επίσης ασχολούμαστε με πολλά προγράμματα που και στο σχεδιασμό είναι πιο φιλοπεριβαλλοντικά και φυσικά μας ενδιαφέρουν και οι λύσεις στο τέλος, αποτελεσματικότητα δηλαδή. Και τελευταίο παράδειγμα, ε, νέα παπούτσια χωρίς χρώμιο. Έχουμε ένα βιολογικά παπούτσια. Υπάρχει, νομίζω, πολύ ενδιαφέρον από την αγορά για τέτοιου είδους ε, ε, παπούτσια. <laughs> Ευχαριστώ. Good morning, everybody. Uh, finally, Καλή σας μέρα για την Enterprise Euro Network που έχει ως στόχο να βοηθήσει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την πρόσβασή τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι μάνατζερ των μικρών και μισών επιχειρήσεων δεν έχουν πάντα το χρόνο να αναζητήσουν τη χρηματοδότηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκουν δύσκολο να μεγαλώσουν τι επιχειρήσει του, αντίθετα από τι μεγάλε βέβαια επιχειρήσει. Το ε, δίκτυό μας είναι ένα one-stop shop, μια μοναδική θηρίδα δηλαδή για ό,τι έχει σχέση με τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Ε, ξεκινήσαμε το 2008 και είμαστε αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο δίκτυο όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίω που συνδέει επιχειρήσεις με την Ευρώπη και ε, το αντίθετο βέβαια. Έχουμε περίπου 600 σημεία ε, επαφών σε 49 χώρες, καλύπτουμε βέβαια όλες τις περιφέρειες ε, της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, καθώς και σε στατικές αγορές εκτός της Ένωσης. Περίπου 3.000 εμπειρογνώμονες είναι λοιπόν δίκτυο ανθρώπων που προσφέρουν συμβουλές στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις και δίνουμε πρακτική βοήθεια. Δηλαδή, για παράδειγμα, μεταφράζει δύσκολα νομοθετικά κείμενα σε μια γλώσσα που μπορούν πιο εύκολα να καταλάβουν οι ε, διαχειριστές των μικρών και μεσών επιχειρήσεων αλλά βέβαια κάνει και άλλα πράγματα, όχι μόνο αυτό ε, δημιουργεί ευκαιρίες για business και βρίσκει επαφές με άλλους ε, εταίρους επιχειρήσεων και γι' αυτό διατηρεί μια τράπεζα δεδομένων για παράδειγμα για την μεταφορά τεχνολογίας η μεγαλύτερη τράπεζα δεδομένων με 13.000 προφίλ προσφορών τεχνολογίας αλλά και ζήτησης. Το άλλο ε, που κάνουμε είναι να ακούμε τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, όπως είπε ο διευθυντής μου προηγουμένως, το δίκτυο δίνει feedback του τι πετυχαίνει και του τι δεν πετυχαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι μία από τις πηγές που στην βάση τους μπορούν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κρίνουν αν μία πολιτική συγκεκριμένη λειτουργεί ή όχι, αποδίδει ή όχι. Και το δίκτυο είναι ένα καλό παράδειγμα μιας κοινοπραξίας ε, στην βάση της επικουρικότητας, άρα δεν χρειάστηκε να επανεφεύρουμε τον τροχό, ας το πω έτσι, και γι' αυτό τα γραφεία μας φιλοξενούνται ε, σε σημαντικές οργανώσεις όπως για παράδειγμα εμπορικά επιμελητήρια, ε, οργανισμούς που προωθούν την ανάπτυξη, πανεπιστήμια, τεχνολογικά ιδρύματα και ούτω που όχι μόνο μας φιλοξενούν, αλλά συμβάλλουν και σημαντικά και χρηματοδοτικά στην επιτυχία του δικτύου μας. Και ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ επιτυχημένη η φόρμουλα αυτή. Σε ό,τι αφορά ποσοτικά αποτελέσματα, έχουμε καταφέρει τα τρία πρώτα χρόνια να φτάσουμε, να προσεγγίσουμε 2,5 εκατομμύρια μικρές και μεσές επιχειρήσεις, σε διαφορετικά επίπεδα βέβαια. Συνολικά 20.000 εκδηλώσεις έχουμε διοργανώσει και έχουμε έτσι προσκαλέσει το ενδιαφέρον 750.000 μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 66.000 εταιρείε έχουν έλθει σε ε, ε, εκδηλώσεις για διαμεσολάβηση, όπου μπορούν να βρουν δηλαδή ε, τρόπο επαφής με άλλες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αναπτύξουν το χαρτοφυλάκιό τους. Το δίκτυό μας βοηθεί επίσης μικρές και μεσές επιχειρήσεις για να εξεύρουν χρηματοδότηση από το, από το, πρόγραμμα, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα 7, ε, για την έρευνα δηλαδή, και σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματά μας έγινε μια ε, επιθεώρηση πέρσι και είδαμε ότι πάνω από τις μισές εταιρείες οι οποίες προσήλθαν σε εκδηλώσεις μας απέκτησαν πρόσβαση σε νέες αγορές ε, πάλι περίπου οι μισές ή και λίγο παραπάνω έχουν αναπτύξει ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία ε, επίπτωση στις, ε, στον, στον τζίρο τους είχαν πάλι 50% 40 από αυτές έχουν βελτιώσει έχουν, 45% έχουν βελτιώσει τεχνολογία του, 40% έχουν αρχίσει ένα καινούριο business project και 99,7% των επιχειρήσεων αυτών θα συνιστούσαν τις υπηρεσίες μας σε άλλους. Έχουμε βέβαια και άλλε ε, ιστορίε επιτυχία από τη Γερμανία και την Ιταλία, εκεί στο πίσω μέρο τη αίθουσα που μπορείτε να τα βρείτε, ε, για την, ε, μια επιχείρηση που λέγεται Leva και είναι από το Leverkusen και που ασχολείται με την αφαίρεση επικίνδυνων ουσιών από βιομηχανικά απόβλητα. Και αυτοί έψαχναν να βρουν νέε αγορέ. Του φέραμε σε μια εξειδικευμένη έκθεση και βρήκαν έναν άλλο επιχειρηματία στην Ιταλία που ήταν διατεθειμένος να περιλάβει την τεχνολογία αυτή στο χαρτοφυλάκιό του. Χαρτοφυλάκιο του επομένω ήταν μια επιτυχία και για τις δύο αυτές πλευρές. Το άλλο παράδειγμα είναι από την Δανία και το Ενωμένο Βασίλειο η επιχείρηση, μια εταιρεία μάλλον που λέγεται APRO και η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή ε, ανεμογεννητριών που τοποθετούνται ε, μακριά από την ακτή και αναζητούσε καθώς επίσης και μια δανική ε, επιχείρηση ε, επαφή με, ε, με πιθανούς εταίρους έκαναν λοιπόν μια κοινοπραξία και αυτή κατέληξε εν τέλει στην πρόσληψη 30 εργαζομένων και στις δύο χώρες δηλαδή δημιουργήθηκαν 30 θέσεις εργασίας αυτά είναι ολίγες και σας ευχαριστώ ο Πρόεδρος ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι για την πλήρη ενημέρωση. Έχουμε τώρα τους πρώτους συναδέλφους, τέσσερις στον αριθμό που ζητούν το λόγο. Υπάρχει κανείς ακόμη. Τότε μπορώ να κλείσω τον κατάλογο. Α, βλέπω τον κύριο Ρούμπικ. Για μετρήστε παρακαλώ. Ναι, ναι, σας έχουμε, σας έχουμε σημειώσει. Έξι λοιπόν. Αν θέλουμε να μπορέσουν να μας απαντήσουν οι, οι δήμονες θα πρέπει να περιοριστείτε σε δύο λεπτά. Δεν βλέπω άλλο τρόπο. Κύριε Καρβάλιο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λαμπέρ και τους συνεργάτες του από, την, από τον οργανισμό ΕΑΣΥ, τον εκτελεστικό οργανισμό καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας. Παρακολουθώ το έργο σας εδώ και πολλά χρόνια, κυρίως από την προηγούμενη μου ιδιότητα ως πανεπιστημιακού, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζω τα προγράμματα ε, και εντυπωσιάστηκα και από την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των, της διαχείρισης των προγραμμάτων σας, αλλά και από την εύστοχη επιλογή αυτών των προγραμμάτων. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων ε, θα έχουν μεγάλη σημασία για την υλοποίηση και των διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων και θα βοηθήσουν την εφαρμογή των πολιτικών, την διάδοση των καλύτερων πρακτικών και για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, νομίζω ότι αυτό το δίκτυο με τους δημάρχους είναι πολύ χρήσιμο και μπλέκει γύρω στους 2.000 πόλεις και δημάρχους. Επίσης ε, είναι σημαντικό για την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα, ιδιαίτερα στο αστικό περιβάλλον. Έχω δύο ερωτήσεις. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το μέλλον. Χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε το μελλοντικό προϋπολογισμό με μια αύξηση ε, για τον προϋπολογισμό έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι περιμένετε για τα δικά σας προγράμματα, πώς βλέπετε τον προϋπολογισμό τους, επίσης πώς βλέπετε τη δομή του εκτελεστικού οργανισμού στο πρόγραμμα πλαίσιο. Πιστεύετε ότι υπάρχει περαιτέρω ολοκλήρωση στο μέλλον. Δεύτερη ερώτηση. Στο παρελθόν είχατε ένα πρόγραμμα ε, συνεργασίας με αναπτυσσόμενες χώρες. Τώρα έχει παράσει τη Europaid. Κατά τη γνώμη μου, εσείς διαχειριζόσασταν καλύτερα το πρόγραμμα από τη Europaid γιατί εσείς καταλαβαίνετε καλύτερα την ενέργεια, το θέμα της ενέργειας. Υπάρχει κάποια ε, πιθανότητα να ανακτήσετε τη διαχείριση των προγραμμάτων συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες για θέματα ενέργειας. Ευχαριστώ. Η κυρία Μέρκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές για την παρουσίασή σας. Η φήμη σας έχει φτάσει ως εμάς, προηγείται της παρουσίας σας της φυσικής, από πολλά καλά λόγια και σας ευχαριστώ για τα αποτελέσματα, τα συγκεκριμένα που μας παρουσιάζετε, τα χρειαζόμαστε. Τώρα κάποιες ερωτήσεις ίσως προκλητικές λίγο για την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης really need Europe in uh, ε, Για τον οργανισμό σας, που προέρχεται από τον οργανισμό σας. Προφανώς τα προγράμματα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Γιατί όμως θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκά τα προγράμματα αυτά. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το αν χρειάζεστε μια συνεργασία εταιριών από πολλές χώρες. Γιατί κάποια από τα προγράμματα αυτά ίσως να λειτουργούν καλύτερα αν υποστηρίζονται σε εθνικό επίπεδο. το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Το εμείς θα θέλαμε εδώ κάποια πιο πρακτικά στοιχεία, θα θέλαμε μεγαλύτερη απλοποίηση. Έχουμε πολλές υπηρεσίες εξωτερικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές από αυτές κάνουν εξαιρετική δουλειά. Το θέμα είναι χρειάζονται όμως πράγματι τόσες υπηρεσίες. Μήπως χρειαζόμαστε λιγότερες υπηρεσίες που θα κάνουν ακόμα καλύτερη δουλειά. Πώς συνδυάζεστε σαν παράδειγμα με το πρόγραμμα αέρια. Γιατί και οι δύο απευθύνεστε προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως έχουμε ήδη πει στα πλαίσια των εμβληματικών πρωτοβουλειών για την τεχνολογία, εμείς θέλουμε ε, μία μόνο απευθυντική θηρίδα για την υποδοχή όλων αυτών των προγραμμάτων. Είναι εύκολο να σας βρούνε μεν οι μικρομεσαίες, αλλά αν μπορούν να βρούνε τόσες υπηρεσίες αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Και πώς συνεργάζεστε και με τα εθνικά σημεία επαφής. Σε αυτή τη ζούγκλα γενικά διασύνδεσης των ευρωπαϊκών δικτύων. Πώς θα βελτιώσετε ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες σας στα πλαίσια των δικτύων. Ευχαριστώ Τόμας. για τους συναδέλφους. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι η υπηρεσία αυτή είναι το αποτέλεσμα δύο βασικών πολιτικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το 2000 και μάλιστα μετά από μια διακομματική πρωτοβουλία ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργηθεί μια εκτελεστική τέτοια υπηρεσία για την έξυπνη, την ευφυά Ευρώπη και να επικοινωνεί έτσι με τον υπόλοιπο κόσμο. Και επίσης το 2005 ο κύριος Βακάλης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με την έκθεσή του έφερε σε συνεργασία τα προγράμματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν το μωρό αυτό είναι δικό μας. Βέβαια δεν το λέγουν οι υπάλληλοι ε, αυτοί και πρέπει εμείς να το πούμε. Απειλείται γιατί στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο τι θα συμβεί. Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος η υπηρεσία αυτή οι οποίες είναι από τις καθοδηγητικές γενικά υπηρεσίες θα διαιρεθεί από ό,τι φαίνεται και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να καταστραφεί σε αυτό το παιχνίδι πολιτικής που γίνεται ανάμεσα σε ορισμένους επιτρόπους οι οποίοι αναζητούν να ελέγξουν κάποιους τομείς. Είναι λοιπόν σαφέστατο καθήκον της Επιτροπής μας, της Επιτροπής που ασχολείται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, της Επιτροπής η οποία θέλει να προχωρήσει η Ευρώπη στον τομέα των μικρομεσαίων και της καινοτομίας. Πρέπει να είμαι λοιπόν, να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για το τι θέλουν να κάνουν οι μάγοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία ερώτηση για τον κύριο Σατάφ μάλλον. Χάρηκα όταν είδα πόσο σφαιρικό το δίκτυο των επιχειρήσεων ε, είναι. Είστε στη ΣΥΠΑ, στην Κίνα, στη Ρωσία κτλ. Για τις χώρες του Μαγκρέμπ, ένα παράδειγμα. Μήπως έχουμε τώρα μια μεγάλη ευκαιρία να βάλουμε μέσα χώρες όπως η Τινησία, το Μαρόκο, η Αίγυπτος ή και μακράν αυτών η και μακραν αυτον έτσι ώστε να έχουμε έναν ζωντανό τομέα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για το θέμα αυτό στην πολιτική γειτονίας. Σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση και από τα τέσσερα μέλη του οργανισμού. Εγώ δεν γνώριζα όλα αυτά τα προγράμματα και με εκτίμησα ιδιαίτερα σε αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε. Έχω μερικές ερωτήσεις. Οι συνάδελφοι ε, ρώτησαν για τις τρίτες χώρες, αλλά τα προγράμματα αυτά είναι κυρίως ευρωπαϊκά. Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια για την δίκαιη ή ίσως άδικη γεωγραφική κατανομή σε ό,τι αφορά την ε, εκταμίευση κονδυλίων από τα προγράμματα αυτά. Γιατί φαίνεται ότι μερικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι επιτυχείς, αλλά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις από ορισμένες κοινωτικές χώρες είναι απούσες, είναι λιγότερο επιτυχείς. Αυτό που είναι σημαντικό για, το, για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα είναι η εκπαίδευση, η παιδεία. Είναι δύσκολο μερικές φορές να βρούμε μορφωμένους ανθρώπους υψηλής κατάρτισης. Πώς ε, ε συνεργάζεστε με τα διάφορα Ινστιτούτα Καινοτομίας. Ε, αναφερθήκατε στο 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά δεν μιλήσατε για το Ινστιτούτο Καινοτομίας. Στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο Ίσως θα έπρεπε να έχουμε ένα σωστό σύνδεσμο μεταξύ τεχνολογιών, επικοινωνιών και πληροφορίας ε, και προγράμματος ε, πρωτοβουλίας ε, και προγράμματος καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ θερμά τους προσκεκλημένους μας, να τους ευχαριστήσω για τις εξηγήσει και να τους διαβεβαιώσω ότι εμείς ανέκαθεν ήμασταν υπέρ του προγράμματος καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας και ταχθήκαμε υπέρ της χρηματοδότησης. Μάλιστα καταψηφίσαμε μια πρόταση που δεν θεωρούσαμε σωστή για το θέμα αυτό. Μας δώσετε καταπληκτικές εξηγήσει. το έργο σας φαίνεται αξιόλογο, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν και αρνητικές πτυχές. Πείτε μας λοιπόν τι προβλήματα αντιμετωπίσατε και τι πιστεύετε θα πρέπει να αλλάξει στο μέλλον, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να σας βοηθήσουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω μια ερώτηση επίσης για το μέλλον, γιατί εδώ και δύο, λίγο καιρό έχει εξεταστεί η πρόταση να συγχωνευτούν τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας σε ένα ενιαίο πρόγραμμα πλαίσιο. Ποια είναι η δική σας γνώμη, γιατί ξέρουμε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά εσείς που είστε διαχειριστές των βασικών προγραμμάτων για την καινοτομία, τι γνώμη έχετε. Διάβασα και την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος ε, καινοτομίας και θα ήθελα τη γνώμη σας για μία από τις συστάσεις που προτείνει ένα τμήμα της χρηματοδότησης του προγράμματος να χρησιμοποιηθεί για προγράμματα που εμπίπτουν στις ε, προτεραιότητες όπως συνέβη και με το 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο. Για παράδειγμα, μέλλον και νέες τεχνολογίες. Γιατί δεν μπορούμε από την αρχή να προβλέψουμε όλα τα προγράμματα που θα ανακύψουν ή τα προβλήματα που θα ανακύψουμε σε μία επταετία. Άλλωστε η καινοτομία προχωρά με ραγδαίου ρυθμούς. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί αυτή η ευελιξία. Είχαμε αυτή τη σύσταση για το 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο. Εσείς πώς την κρίνετε. Ευχαριστώ κυρία Τωρέα. Και από δική μου πλευρά θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις δραστηριότητές σας τις οποίες γνωρίζουμε. Μια αξιολόγηση η οποία συνδέεται θα έλεγα με τις ανησυχίες που ακούσατε από τους συναδέλφους εμείς δεν θεωρούμε ότι το σύνολο των υπηρεσιών αυτών που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίνεται στο ίδιο σύνολο απαιτήσεων και γι' αυτό στρέφουμε την προσοχή μας θετικά στις εργασίες σας. Δύο σημεία να υπογραμμίσω. Είναι όλο και πιο σημαντικό να μπλουτίσουμε και να υπογραμμίσουμε και να καταστήσουμε τη δραστηριότητά σας ιδιαίτερα αποτελεσματική. Γιατί στρεφόμεθα πράγματι και επιμένουμε για την καινοτομία, την έρευνα και την ενοτομία και όχι την έρευνα εναντίον της καινοτομίας. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να ζητήσω πάρα πολύ γρήγορα να μας δώσετε ένα feedback της δραστηριότητάς σας. Πώς εφαρμόζετε εσείς τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι επιπλέον προσθέτετε εσείς στις ε, συγκεκριμένες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, υπάρχει ένα πρόβλημα για περισσότερα χρήματα, καλύτερη ενημέρωση, απλούστερη λειτουργία τεχνική. Όλα αυτά είναι θέματα στα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε. Ένα δεύτερο θέμα, η πρόσβαση των μικρομεσαίων σε τέτοιου είδους προγράμματα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχει μόνο μία ζούγκλα θεμάτων, αλλά και μία ζούγκλα θα έλεγα προγραμμάτων και διαδρομών για να φτάσει κανείς εκεί. Πώς μπορούμε να απλοποιήσουμε την πρόσβαση αυτή. Πώς μπορούμε να καταστήσουμε την θύρα αυτή, την φιλόξενη, ελκυστική γιατί τότε μόνο θα αυξήσουμε τις πιθανότητες να ωφεληθούν οι μικρομεσαίες. Πώς μπορείτε λοιπόν να καταστήσετε την πρόσβαση των μικρομεσαίων πιο εύκολη. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στους προσκεκλημένους μας που δυστυχώς έχουν μόνο ένα δεκάλεπτο για να απαντήσουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους ευρωβουλευτές, τα μέλη της Επιτροπής για το ζωηρό ενδιαφέρον που έδειξαν για τις παρουσιάσεις που κάναμε από τον εκτελεστικό μας οργανισμό και για τα προγράμματα. Εκτιμούμε ιδιαίτερο αυτό το ενδιαφέρον. Θα προσπαθήσω να απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ερωτήσεις. Ορισμένες αφορούσαν τη συζήτηση που γίνεται στην Επιτροπή και είναι κάπως δύσκολο να απαντήσω γιατί εμεί είμαστε εκτελεστικός οργανισμό. Εκτελούμε τα προγράμματα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο όνομα τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρωταρχικός μας ρόλος δεν είναι η συμμετοχή στη συζήτηση για την διάρθρωση του μελλοντικού πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Τώρα, ποιε είναι οι προσδοκίε μα για το μέλλον. Εμείς παρακολουθούμε προσεκτικά τις συζητήσεις και τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είδαμε τις χθεσινές προτάσεις για το μελλοντικό προϋπολογισμό και διαπιστώνουμε ότι θα έχουμε ένα ξεχωριστό μηχανισμό. Θα πρέπει να το ελέγξω βέβαια, αλλά μάλλον θα υπάρξει ένα ξεχωριστό εργαλείο για την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα δούμε τι σχέση θα διαμορφωθεί μεταξύ αυτού του νέου μηχανισμού και του CSF. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εφής Ευρώπη, ε, ένα τμήμα ε, αναπτυξιακής συνεργασίας με αναπτυσσόμενες χώρες σε θέματα ενέργειας εκχωρήθηκε στην Γενική Διεύθυνση για την Ανάπτυξη, στο EuroPaid μάλλον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα ανάκτηση αυτού του προγράμματος ε, για την ενέργεια και συνεργασία για θέματα ενέργειας σε αναπτυσσόμενες χώρες στα γίνει από εμά. Τα προγράμματα, τα διάφορα αυτά προγράμματα, όπως σας είπα, έχουν μια ορατή ευρωπαϊκή διάσταση και σε ορισμένε περιπτώσεις το απαιτούμε αυτό. Απαιτούμε, για παράδειγμα, τρεις ε, συμβαλόμενους από τρεις διαφορετικές χώρες μέλη. Βέβαια, τα κράτη-μέλη έχουν και τα εθνικά τους προγράμματα. Και είναι σημαντικό εμείς να μπορούμε να αποδείξουμε αυτή την ευρωπαϊκή υπεραξία στα δικά μας προγράμματα, ώστε πραγματικά να γίνει κοινή χρήση της εμπειρογνωμοσύνης και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και της τεχνογνωσίας σε όλη την Ευρώπη. Αυτή είναι η πεμπτουσία της ευρωπαϊκής διάστασης. Ο, σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς, αν θα πρέπει να έχουμε περισσότερους ή λιγότερους οργανισμούς. Και αυτή την ερώτηση θα πρέπει να την απευθύνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τη συζητήσετε μεταξύ σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρία Μέρκης, αναφερθήκατε στη σχέση μεταξύ του δικού μας οργανισμού και του REA. Ε, τώρα έχουμε κοινό κτίριο με τους συναδέλφους από την REA και συγκρίνουμε αυτά που κάνουμε εμείς ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αυτά που κάνουν οι συνάδελφοι προκειμένου να δημιουργήσουμε καλύτερες συνέργειες. Πάντως θα έχουμε στενή συνεργασία στο άμεσο μέλλον και σίγουρα στα πλαίσια των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών. Σημείωσα τα σχόλια του κύριου Τούρμες και χαίρομαι που και εσείς και οι συναδελφοί σας ε, ε, αισθάνεστε την συμπάθεια και την προσήλωση στην, ε, στον οργανισμό μας. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους αργότερα για να απαντήσω σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για το δίκτυο. Η κυρία Σιζέλ είπε ότι φοβάται ότι δεν γίνεται δίκαιη κατανομή των προγραμμάτων μεταξύ των κρατών μελών. Δεν συμφωνώ, γιατί τα προγράμματά μας είναι ανοιχτά σε συμμετοχή προς όλες τις χώρες μέλη. Και το Ευρωπαϊκό Δικτύο για τις Επιχειρήσεις έχει 600 εταίρους σε όλες τις ε, ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο σε ευρωπαϊκές. Εμεί δεν είχαμε τέτοια εμπειρία. Δεν νομίζω ότι τα προγράμματα αυτά αποσιάζουν ε, από ορισμένε χώρες μέλη. Πιστεύω ότι υπάρχει μια δίκαιη κατανομή και ισορροπημένη. Και ίσως το τελευταίο θέμα που θέξατε μπορούμε να το συζητήσουμε και διμερώς. Κυρία Ριέρα Μαντουρέλ, ρωτήσατε αν υπάρχουν και αρνητικές πτυχές, αρνητικές εμπειρίες. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί σε τέτοιου παρουσιάσει εμένουμε στα θετικά στοιχεία και στι θετικέ εμπειρίε. Ίσως στο μέλλον θα πρέπει να επιτείνουμε την απλούστευση και το streamlining. Δεν λέω ότι όλα είναι ρόδινα και τέλεια, αυτό δεν θα ήταν και πολύ ρεαλιστικό, αλλά στο μέλλον που θα έχουμε το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, σίγουρα θα υπάρξει μια περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών μας, ιδιαίτερα χάρη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μας. Εμείς και στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα θέλαμε ο οργανισμός μας να αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα και ένα ε, συνεκτικό πλέγμα καθηκόντων και όχι μόνο ad hoc αποστολές. Σήμερα το πρωί δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε στο μέλλον να έχουμε και ένα ειδικό οργανισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από εσά αν θα το το σκόπιμη ιδέα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον αρμόδιο για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων. Ο κ. Χουσέν Σατάφ, μία ερώτηση κάνατε για την σχέση ε, μέσα στο δίκτυο. Πώς δηλαδή δουλεύουμε με τα εθνικά contact points για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Έχουμε μία ομάδα επαφών όπου συμμετέχουν ορισμένοι από τους εταίρους μας, του δικτύου μας δηλαδή, και τα contact points για να εξετάσουν πώ μπορούν να συνεργαστούν. Μια ιδέα για παράδειγμα μπορεί να είναι ότι το δίκτυο προωθεί τον ρόλο των εθνικών contact points, γιατί συνήθω υπάρχει ένα σε κάθε χώρα. Το δίκτυο λοιπόν μπορεί να παίξει καλό ρόλο και στις περιφέρειες. Να δούμε πώς μπορούν να εργαστούν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά. Οι συζητήσει αυτές συνεχίζονται. Για την ερώτησή σας σχετικά με τα σημεία επαφής σε τρίτες χώρες. Έχουμε όντως στην Τινησία και την Αίγυπτο Επίσης στην Ουκρανία που είναι και το πιο πρόσφατο μέλος μας. Βέβαια ένα κέντρο σε κάθε μια από τις χώρες αυτές εφόσον το ιδιαίτερο βάρος το ρίχνουμε στην Ευρώπη. Θα συναντηθούμε μαζί τους την επόμενη εβδομάδα, έρχονται εδώ και θα δούμε πώς μπορούμε να τους υποστηρίξουμε, να παίξουν ένα ρόλο ίσως για να αναπτύξουν τον ιδιωτικό τομέα, να κάνουν το business development δηλαδή, Προσπαθούμε να τους ε, στηρίξουμε, δεν τους χρηματοδοτούμε όμως, άρα ο ρόλος μας είναι περιορισμένος. Προσπαθούμε κυρίως να τους διασυνδέσουμε με τους εταίρους του δικτύου και τους θεσμούς εδώ στην Ευρώπη. Έτσι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ενισχύσουμε, μπορούμε να στηρίξουμε τις κινήσεις αυτές στις ε, χώρες που προανέφερα. Αν έχετε όμως ιδέες, ασφαλώς θα τις ακούσουμε για τις διαφορετικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και από διαφορετικές χώρες. Για το δίκτυο αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όντως οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Στις νέες χώρες μέλη, αν μπορούμε ακόμη να το πούμε αυτό, υπάρχει ακόμα κενό ενημέρωσης το οποίο πρέπει να καλυφθεί. Ενώ στις παλαιότερες χώρες μέλη περισσότερο υπάρχει, λόγο, υπάρχει ανάγκη τώρα ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Υπάρχει λοιπόν μια μετακίνηση, αλλά βλέπουμε όλο και περισσότερο την ανάγκη αναζήτησης ε, ευκαιριών για επιχειρηματική ανάπτυξη. Και εκεί το δίκτυο μπορεί να παίξει πραγματικά σημαντικό ρόλο. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λάμπερτ, κυρίες και κύριοι, για την ενημέρωση, για την πλήρη απάντηση των ερωτήσεων. Βρίσκω ότι ήταν σημαντικό που ακούσαμε την ενημέρωση αυτή σήμερα και ιδίως εν ώψη των συζητήσεων που ήδη ε, διεξάγονται αλλά και αυτών που θα έρθουν. Θα προχωρήσουμε αμέσως στην ψηφοφορία τώρα. Κυρίε και κύριοι, θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, αγαπητέ και αγαπητοί συνάδελφοι. Ελπίζω ότι είστε όλοι παρούσε ή παρόντε, αναλόγω, και ελπίζω ότι έχετε τι ηλεκτρονικέ σα κάρτε. Θέλετε να δοκιμάσουμε αν λειτουργεί, να, να κάνουμε μια δοκιμή, αν λειτουργεί ε, σωστά το σύστημα. Wir versuchen einmal die Abstimmung θα κάνουμε μια πρώτη δοκιμή, αν θέλετε. Ποιος θεωρεί ότι αύριο θα είμαστε όλοι ακριβείς στην ώρα μας. Αυτό θα, θα βάλουμε ως θέμα ψηφοφορίας. Πέρας, το αποτέλεσμα είναι... Α, δεν βλέπουν διερμηνείς το αποτέλεσμα, τώρα το βλέπουν 26 Υπέρ 6 κατά. Μάλιστα. Ποιοι είναι αυτοί οι 6. Καλά, καλά. Αρχίζουμε λοιπόν. Έχουμε ορισμένες ψηφοφορίες, τις οποίες θα πρέπει να διεξαγάγουμε. Σας παρακαλώ, ακούστε με για λίγο. Καλύτερα θα είναι, θα είναι πιο εύκολα. Θέλω να πω μια φράση. Έχουμε μια εκτεταμένη ψηφοφορία για την έκθεση για τις πρώτες ύλες. Εχθές το βράδυ στις 9 έλαβα την λίστα ψηφοφορίας για την ψηφοφορία αυτή. Έχουμε βέβαια ένα σχέδιο, ένα πλάνο για το πώ ε, φτιάχνουμε τι λύσει ψηφοφορία. Ορισμένε φορέ επιτυχαίνει, ορισμένε φορέ όχι. Για την επόμενη ψηφοφορία, εφόσον φτάσει η λίστα τόσο αργά και οι συνάδελφοί μου δεν έχουν τη δυνατότητα να την εξετάσουν, τότε δεν θα ψηφίσω. Και ούτε καν θα το συζητήσουμε. Θα είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτά ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να βγάλω από το στήθο μου. Ερχόμαστε τώρα στο 4, δηλαδή τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση τη κοινή επιχείρηση Κυψέλε Καυσίμου και Ιδρογόνου συμφωνήσαμε απλουστευμένη διαδικασία στους συντονιστές και επειδή κανείς δεν έχει προβάλει ενστάσεις θεωρώ ότι μπορεί να εγκριθεί. Και προχωρούμε στο επόμενο, δηλαδή στο υπαριθμό 5, με συγχωρείτε, ο κύριος Τούρμες. Εμείς είχαμε σκοπό να απόσχουμε, όχι διότι δεν θεωρούμε σημαντική τεχνολογία της κυψέλες ε, καυσίμου, αλλά διότι θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας λέει ολόκληρη την αλήθεια σχετικά με το πόσο καλά λειτουργεί ή πόσο δεν λειτουργεί αυτή η κοινοπραξία, αυτό το joint venture. Γι' αυτό θέλουμε μετά το καλοκαίρι να γίνει προσπάθεια να κατανοήσουμε πώς καλό λειτουργεί, διότι οι πληροφορίε που έχουμε είναι ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όσο μας τα παρουσιάζουν. Φαίνεται πως έχει πληροφορίε από την Κομισιόν που δεν έχουν άλλοι. Πάντως αυτό που λες πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ναι, ε, στην περίπτωση αυτή μπορεί και να αναβληθεί μια ψηφοφορία για να διευκρινιστεί το θέμα. Τέλο πάντων, τώρα πάντω εγκρίθηκε. Όπω είπα, το 5. Μέθοδη πρόσβαση στην κυβερνητική υπηρεσία που προσφέρεται από το Παγκόσμιο Σύστημα Δορυφορική Ραδιοπλοήγηση που προέκυψε από το πρόγραμμα Γαλιλαίο. Εδώ έχουν διεξαχθεί διαπραγματεύσει, συζητήσει. Έχει γίνει πολλή δουλειά. Δυστυχώ ο κύριο Γκλάντε δεν είναι παρόν, ο οποίο δούλεψε πολύ για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ψηφίσουμε τώρα το συμβιβαστικό κείμενο. Ποιος ψηφίζει υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αποχές. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία αυτή πρέπει να γίνει με ονομαστική ψηφοφορία, δηλαδή ηλεκτρονική. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Μα τι συμβαίνει, κύριε 38 υπέρ 4 κατά. Εγκρίθηκε. Για να σας θυμίσω ότι δεν έχω την κάρτα και γι' αυτό ψηφίζω δια ανατάσεως της χειρός. Ο πρόεδρος, καλά, λείπει μια κάρτα. Παρέμβαση της κυρίας Εκ χωρίς μικρόφωνο. Ο κ. Παναγιωτόφ ψηφίζει αλλά δεν έχει την κάρτα του. Α, μάλιστα, δεύτερη κάρτα που λείπει λοιπόν. Σεις επίσης δεν λειτουργεί το μηχάνημά μου, αλλά ίσως να μην πάτησα σωστά το κουμπί. Καλά, ούτε και εγώ μπορώ να το ξέρω βέβαια αυτό. Δεν μπορώ να απαντήσω σε τέτοια τεχνικά θέματα. Αλλά πάντως σας ευχαριστώ για την ε, υπόδειξή σας. Τα σημειώσαμε όλα αυτά. Ερχόμαστε στο ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου που επίσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Θα ε, κάνουμε δοκιμή αν λειτουργεί τώρα πάλι το μηχάνημα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. ...37 υπέρ, 3 κατά και 4 αποχές. Εσείς ήσασταν υπέρ που δεν έχετε την κάρτα σας. 38 λοιπόν. Κύριε Παναγιώτοφ, υπέρ. Υπέρ επίσης. 39 υπέρ, 3 κατά, 4 αποχές εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ όλες και όλους όσοι κατέβαλαν σχετικές προσπάθειες. Ερχόμαστε τώρα στην έκθεση πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες την οποία έχει συντάξει ο κύριος Μπιουτικόφερ με συνεργασία άλλων. Υπάρχουν και πολλές συμβαστικές τροπολογίες, ευτυχώς. Θα αρχίσουμε. Πρέπει να αλλάξει κάποιος. Αρχίζουμε με την συμβαστική υπαριθμών 2, αν, αν ε, Μα δεν είναι, δεν είναι και λογικό, δεν είναι και λογικό. Μάλλον θα προαρχίσω με την υπαριθμόν 1. Αυτό συμβαίνει και συνήθως. Σας ευχαριστώ που μου το υποδείξατε. Συμβαστική 1 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 3α υπέρ παράγραφος 3α συγγνώμη παράγραφος 3α αλλά συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 120 υπέρ Κατά. Α, ας, ας επαναλάβουμε. Ή μάλλον όχι, θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει. Πέρας. Και απερίφθη. Α, ναι, συγγνώμη, υπάρχουν και ορισμένοι χωρίς, χωρίς κάρτες. Πώς ψηφίζετε. Κατά. Και εσείς κύριε Παναγιώτοφ. Υπέρ ή κατά. Κατά. Απορρίπτεται επομένω. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 17 υπέρ θέλετε επαλήθευση της 152 152 επαλήθευση αλλά νομίζω ότι ήταν σαφές καλά λοιπόν η ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρας και απερίφθη συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή συμβαστική 19α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 181 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος, επαλήθευση δηλαδή. 181, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 183 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 185 σε τρία τμήματα. Πρώτο, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. Τρίτο τμήμα, επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίθηκε. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Συγγνώμη, 194 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. 194. Επαλήθευση αρχίζει. Πέρας. Και εγκρίθηκε. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 225 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 200... Τη 225 θέλετε. Επαλήθευση. Με ηλεκτρονική ψήφο. Πέρας, ψηφίστη, υπερψηφίστηκε. 208 σε δύο, σε δύο τμήματα. Α, μόνο το δεύτερο μέρος. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 224 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 230 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 231 σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά επαλήθευση επαλήθευση του δεύτερου τμήματος αρχίζει πέρας απερίφθη 235 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 257 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται 240 υπέρ θέλετε επαλήθευση 257 αρχίζει Πέρασε. Απέριφθη. 240 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 241 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 251 σε τμήματα. Μόνο το δεύτερο τμήμα. Έτσι δεν είναι. μόνο το τρίτο μέρος, όχι το δεύτερο, το δεύτερο. Το δεύτερο. Λοιπόν, 251, το δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Δεύτερο μέρος υπέρ. Συγγνώμη, τρίτο μέρος λέει πρόεδρος. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 255 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 256 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 258 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 265 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εγκρίνεται εγκρίνεται διόρθωνη πρόεδρος βεβαίως το συμβαστή 29 υπέρ. Ο κύριος Τούρμες επιπλήττει τον πρόεδρο. Συμβαστική 29 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε στα περίφημα recital τις αιτιολογικές σκέψεις. Ε, τροπολογία 8. Με προφορική τροπολογία, ναι. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 9. Με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. αποχέ. εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 12. Με κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Μ, ας επαληθεύσουμε δεύτερο τμήμα λοιπόν επαλήθευση πέρας εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 Α, όχι, ναι, ναι, εκπίπτει αυτή. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πω, πω, πω, όλα του κύριου Μπιτικόφερ, λέει ο πρόεδρος. 25 Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 με προφορική τροπολογία παρακαλώ. 22, 22 λοιπόν υπέρ. Είναι πολύ αργά τώρα κύριε Μπιτικόφερ. Υπέρ λοιπόν τη 22. 22, 22 υπέρ. Κατά. Κατά, όπως είπα, παρακαλώ η κατά, ψήφι κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3, 4, 5 3, 4, 5 όλα μαζί 3, 4 και 6 λέει ο κ. Μπιτικόφερ 3, 4, 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται ερχόμαστε στο recital C υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπάρχουν και γνωμοδοτήσεις 19 14 14 πρώτα, έτσι δεν είναι. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Της ε, Επιτροπής Αναπτύξεως, 6 πρώτα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτή. 11, πάντα της ΔΕΒΕ, πρώτο, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13, α, το πρώτο εκπίπτει, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και προχωρώ στην 18. Δεύτερο τμήμα υπέρ με προφορική τροπολογία υπέρ όπως είπα κατά αποχές εγκρίνεται 30 τώρα α 20 20 συγγνώμη λέει ο πρόεδρος 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το πρώτο τμήμα αυτό δεύτερο τμήμα τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 σε δύο τμήματα μόνο το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται στην Επιτροπή Ιντα εδώ τα πράγματα είναι λίγο συγκεκριμένα παράγραφος 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 πάλι το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 το πρώτο τμήμα εκπίπτει το δεύτερο με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 σε δύο τμήματα Πρώτο, υπέρ. Κατά, είπε ο πρόεδρος, ναι. Την πατήσατε, κατά. Τώρα όχι λέει στο 15, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 16 πρώτο μέρος. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται περιβάλλοντος Τέσσερα. Μόνο το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. πέντε υπέρ κατά επαλήθευση με ηλεκτρονική ψήφο. Πέρας. Εγκρίθηκε. Και οι δύο χωρίς κάρτες είστε υπέρ ή κατά. Είστε κατά. Α, καλά τότε. Δεν, δεν ακούμε δυστυχώς, δεν υπάρχει μικρόφωνο. Α, έχετε την κάρτα σας τώρα. Α, καλά λοιπόν. Η 7 υπέρ κατά απορρίφθηκε. 10. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Α, εγκρίνεται, συγγνώμη. Ε, σαφ, σαφώς. 14 υπέρ. 14. 14 πρέπει να ψηφιστεί. Υπέρ της 14, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18. Η πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ κατά αποχές οι σοσιαλιστές παρακαλώ. Ναι ή όχι. Α, σηκώστε τα χέρια σας καλά γιατί αλλιώ θα νομίζω ότι δεν είστε στην αίθουσα. Απερίφθη λοιπόν. Εγκρίθηκε λέγουν κάποιοι δίπλα του. Ας το επαναλάβουμε. Υπέρ. Μάλιστα εγκρίθηκε. 22 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 24 Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Θα... Υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Υπάρχει ένσταση κατά αυτής. Ο κ. Μπιουτικόφερ ενίσταται. Μέχρι τώρα τι είχαμε δεχτεί όλες τις προφορικές τροπολογίες. Αν όμως υπάρχει έστω και μια, ε, και ένσταση, ε, είναι, δεν είναι παραδεκτή. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο. Η 24 λοιπόν χωρί την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Ε, 28. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται γεωργική μα όλες οι επιτροπές κατέθεσαν μαζί σχεδόν όλες τρομερό θα πρέπει να γράψουμε επιστολή στην Επιτροπή η οποία δεν συνεργάστηκε μαζί μας γιατί αρνεί το καθήκον τη. Τέλο πάντων, παράγραφο 1. Υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. 2 υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. 3 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, οκ, okay, 3 υπέρ, 3 υπέρ, κατά. Θέλετε επαλήθευση. Καλά, καλά λοιπόν. 3 αρχίζει. Πέρας. Ναι. Βλέπετε το αποτέλεσμα. Ε, τέσσερα. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έξι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εφτά υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οχτώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εννέα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ας επαναλάβουμε. 17 υπέρ. 17 υπέρ. Κατά. Ναι, ναι, σαφές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 σε δύο τμήματα. Πρώτο ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αυτό. Τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Και. Α, εγκρίθηκε η έκθεση. Συγχαρητήρια λοιπόν. Και εσείς ήσασταν υπέρ κυρία, έτσι είναι. κυρία τώρα. Ε, ο κύριος Ρούμπιχ θέλει να προβεί σε δήλωση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συγχαρώ τον κύριο Μπιούτι Κόφερ, διότι οι διαπραγματεύσεις ήταν δυσχερείς. Τις διεξήγαγε όμως με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο και για το μεγαλύτερο μέρος της εκθέσεως επειδή είχαμε ε, καλές συμβαστικές τροπολογίες. Ωστόσο θέλω να διαμαρτυρηθώ και θέλω να εγγραφεί στα πρακτικά θέλω να εγγραφεί στα πρακτικά, επαναλαμβάνω, ότι από έξω από το κοινοβούλιο δραστηριοποιούνται λόμπι και μάλιστα προβαίνουν σε προσωπική δυσφήμιση ευρωβουλευτών και μάλιστα ε, μέλη λόμπι τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο μητρό των ε, λόμπιστς του Κοινοβουλίου. Και γι' αυτό ζητώ ε, να σημειωθεί και να υποβληθεί στον ε, γραμματέα του Κοινοβουλίου, διότι τέτοια πράγματα είναι απολύτως απαράδεκτα. Πρόκειται για εκστατεία λάσπης κατά μεμονωμένων ευρωβουλευτών. Αυτό δεν συνάδει προς το κύρος του σώματος. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Βλέπω και από τα χειροκροτήματα των συναδέλφων ότι συμφωνούν. Θα παρακαλέσω τη γραμματεία να το μεταβιβάσει, να το διαβιβάσει μάλλον, συγγνώμη. Και ερχόμαστε στο 7 θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού 2012, όπως σε τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο. Για φανταστείτε ποιος θα πάρει το λόγο, ο κύριος Μπιουτικόφερ. You the floor. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν στις 20 Απριλίου ενέκρινε το σχέδιο προϋπολογισμού και όπως γνωρίζετε προτείνουν αύξηση υποχρεώσεων αλλά και πληρωμών κυρίως επειδή υπάρχουν πολλές εκκρεμείς υποχρεώσεις από παρελθόντα έτη. Η υιοθέτηση του προϋπολογισμού από το Συμβούλιο προβλέπεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα και θα έλθει στο Κοινοβούλιο η πρόταση για τον προϋπολογισμό στο τέλος του μηνός Ιουλίου, 25 Ιουλίου. Στις 11 Ιουλίου ένας τριμερής διάλογος ανάμεσα στην Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα οργανωθεί αλλά εμείς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτόν τον τριμερή διάλογο σε αυτή τη φάση, ίσως αργότερα. Περιμένουμε από το Συμβούλιο να προτείνει μεγάλες ε, μειώσεις στις πιστώσεις πληρωμών στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Η έκθεση Μπαρσάνη, η οποία βρίσκεται στη βάση του συγκεκριμένου τριμερούς διαλόγου, υπογραμμίζει τουλάχιστον σε πέντε επιμέρους σημεία τις θέσεις τις οποίες έχει υποστηρίξει η Επιτροπή μας ιδιαίτερα έντονα στο παρελθόν. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ευγνώμονες στην κυρία Μπαλζάνη που δέχτηκε τις προτάσεις μας και που κατέστησε το θέμα αυτό θέμα όχι μόνο δικό μας αλλά και της Επιτροπής Προϋπολογισμού και της Ολομέλειας η οποία το υπερψήφισε. Είναι εναντίον λοιπόν αυτών των οριζόντιων μειώσεων σε ευρία κλίμακα στον προϋπολογισμό και υπογραμμίζει την ανάγκη να ευθυγραμμιστεί η δημοσιονομική πολιτική με την πολιτική μας στον τομέα της Ευρώπης 2020 και προτείνει επίσης οι αυξήσεις να μην πάνε πέρα από αυτά τα οποία προβλέπουν οι προοπτικές. Προτείνει επίσης το σεβασμό των προτεραιοτήτων για τις αϊφόρες πηγές ενέργειας, όπως επίσης And Επίσης, προτείνει και τη διεύρυνση του ερευνητικού προγράμματος για το 2012-2013. Το Κοινοβούλιο τον Μάιο προετοίμασε μία σειρά προτάσεων για πιλωτικές δράσεις και προπαρασκευαστικές δράσεις και τις έχει ήδη δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αρχίσει να έρχεται την επόμενη εβδομάδα και θα είναι η βάση των αποφάσεων τις οποίες θα πάρουμε εμείς για το ποιες από τις προτάσεις για τα πιλωτικά και τις προπαρασκευαστικές δράσεις που προτάθηκαν από τα μέλη μας θα υποστηριχθούν από το σύνολο της Επιτροπής. Αυτά όλα θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα κατά τη διάρκεια της συνάντησης των σκιωδών εισηγητών. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ. We Όντως βρισκόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή. Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του 2012, εγώ θα προτιμούσα πάγωμα. Η αύξηση 4,1% στις πληρωμές που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε ρεαλιστική είναι ούτε πολιτικός εφικτή στην παρούσα κατάσταση. Βέβαια, θα πρέπει να θέσουμε τις προτεραιότητές μας και να κάνουμε κάποιες προσαρμογές για να προβάλλουμε τις προτεραιότητες και να κρατήσουμε ένα κοινοτικά ουδέτερο προϋπολογισμό. Αν θέλουμε να έχουμε αύξηση δαπανών σε ορισμένου τομεί, θα πρέπει να αφαιρέσουμε από άλλους. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ποια είναι η προτεραιότητά μα και σίγουρα η ενέργεια είναι προτεραιότητα. Εκεί χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια, γιατί όλοι λένε ότι η ενεργειακή πολιτική είναι νευραλγική πολιτική. Ο προπολογισμό ενέργεια για το 2012 προβλέπει μείωση κατά 0,1% και η ενέργεια είναι μόνο μισό τα του συνολικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι είναι σημαντικό το σχέδιο για την ενέργεια, αλλά δεν υπάρχει ξεχωριστή δημοσιονομική γραμμή για το σχέδιο ΣΕΤ. Θέλουμε όμως να χρηματοδοτηθεί το σχέδιο ΣΕΤ. Αυτό είναι πρωταρχική σημασία και για την ανάπτυξη και για την απασχόληση, αλλά και για να εκπληρώσουμε τους περιβαλλοντικούς μας στόχους. Θέλουμε να προωθήσουμε τις νέες τεχνολογίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ΣΕΤ. Πέραν του ε, θέματος ε, της ε, χρηματοδότησης του ΙΤΕΡ, που είναι 1,7 δις ακόμη και να αφήσουμε το ίτερ κατά μέρου, έχουμε τη χρηματοδότηση άλλων ενεργειακών προγραμμάτων που αντιπροσωπεύουν 350 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε μόνο 100 εκατομμύρια ευρώ για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Κάτι πάει στραβά λοιπόν. Υπάρχει ένα γενές λάθος στην ισορροπία αυτού του προϋπολογισμού. Και από τη στιγμή που οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια βρίσκονται στο επίκεντρο των στόχων μα για την υλοποίηση των κλιματικών ε, στόχων που έχουμε, θα πρέπει να αυξήσουμε τα κονδύλια για τις ανανεώσιμες πηγές, αντί να χρηματοδοτούμε άλλους τομείς που δεν αποτελούν προτεραιότητές μας. Ευχαριστώ, δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο. Ε, δεν ξέρω αν θα πρέπει να σας το επισημάνω, αλλά ας το κάνουμε καλύτερα. Έχουμε αυτή τη συνάντηση των σκιωδών για την οποία μίλησα προηγουμένως που θα γίνει στις 7 Εβδόμου. Και εκεί θα ακούσουμε την συζήτηση, μάλλον την άποψη της Κορεπέρ και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα pilot project και τις ε, προπαρασκευαστικές δράσεις και για την κατάθεση τροπολογιών προθεσμία στην Επιτροπή Ήτρε προβλέπεται η 23η Αυγούστου το μεσημέρι. Ε, στην Επιτροπή προπολογισμών που είναι αρμόδια επί η σχετική προθεσμία είναι η 8η Σεπτεμβρίου πάλι το μεσημέρι. Η ψηφοφορία στην Ήτρε θα γίνει στις 30 ε, Αυγούστου και βεβαίως καλούνται τα μέλη να συντάξουν και να καταθέσουν τροπολογίες. Καλά, σας ευχαριστώ. Η κυρία Εκ. Ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο τόσο αργά. Από άψη αρχής είναι σημαντικό να τονίσουμε το ίτερ. Βέβαια έχουμε μια πηγή ενέργειας που είναι η πυρηνική, αλλά θέλουμε να προβλέψουμε χρηματοδότηση για κάτι, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την αντίστοιχη νομοθετική εξουσία, κάτι που δεν ισχύει για το ίτερ. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό με το Συμβουλίο, θα το αφαιρέσουν τελείω ή θα μα εξασφαλίσουν απόφαση και για το πρόγραμμα ίτερ. Ο κ. Ρούμπιχ, ευχαριστώ. Το Κοινοβούλιο έχει ταχθεί εντατικά ή έντονα καλύτερα και υπέρ της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού ε, Τεχνολογικού Ινστιτούτου με ένα πρώτο ποσό τριών δισεκατομμυρίων. Θα πρέπει να εξετάσουμε εάν η προσέγγιση αυτή που θα ωφελήσει τα σχολεία και τα πανεπιστήμια γιατί θα τους προσφέρει πρόσβαση στις πιο πρόσφατες γνώσεις να καταλήξει και μέχρι τους δασκάλους και τους μαθητές για να διασφαλιστεί μια καλύτερη εκπαίδευση που θα ωφελήσει πάλι τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. δηλαδή τα πλονεκτήματα από το 7ο και 8ο προγράμματα πλαίσιο για την έρευνα να καταλήξουν να ωφελήσουν πραγματικά τους ανθρώπους. Α, με συγχωρείτε, ναι, εσείς. Ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν ε, πρόλαβα να πάρω το λόγο πριν δευτερολογήσει ο κύριος Μπιουτικόφερ. Θα είμαι λακωνικός πάντως. Ε, δεν υπάρχει τσεχική διερμηνία ή υπάρχει πρόβλημα στην αγγλική διερμηνία. Θα επαναλάβω. Επαναλαμβάνω, θα είμαι σύντομος. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για την επιχείρηση GSA, για τον οργανισμό, συγγνώμη, GSA. Από ό,τι ξέρω, το Συμβούλιο θέλει να περιορίσει τον προϋπολογισμό για αυτόν τον οργανισμό, κάτι που θα ε, καταστήσει δύσκολο το έργο αυτής της υπηρεσίας της Πράγας. Νομίζω ότι σε ορισμένους τομεί όντω θα πρέπει να κάνουμε κάποιες οικονομίες. Αλλά σε άλλους τομεί θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τι δραστηριότητε, Νομίζω θα πρέπει τον οργανισμό GSA για το Γαλιλαίο να το χρηματοδοτήσουμε. Σα ευχαριστώ. Αν δεν ε, ζητεί κανεί να λάβει το λόγο θα πω τότε ότι έχουμε προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών 23 Αυγούστου και <clears throat> θα προχωρήσω στο επόμενο θέμα της ημερικής διατάξης που είναι το υπαριθμό 8 έλεγχος των κινδύνων που συνδέονται με μείζωνα ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται επικίνδυνες ουσίες. Με εισηγητή τον κύριο Ενά, ο οποίος θα λάβει ω πρώτο τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες οι οποίοι με βοήθησαν στο συγκεκριμένο θέμα και ιδιαίτερα την συνεργάτηδα που είναι δίπλα σας κύριε Πρόεδρε η οποία δούλεψε εξαιρετικά. Λάβαμε υπόψη μας όλα όσα είπαμε και κατά τη διάρκεια των προηγούμενων συναντήσεων. Και συντάξαμε και τροπολογίες που λαμβάνουν υπόψη τους προσανατολισμούς τους οποίους θέλουμε να ακολουθήσουμε. Το ότι δηλαδή υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες χορήγησης εξαιρέσεων, αυτό θα θέλαμε να αλλάξει, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη και η υπεργολαβία σε όλες τις πλευρές και στον τομέα της ασφαλείας. Έτσι οι προθεσμίες θα πρέπει να είναι γραμμένες με συγκεκριμένο τρόπο, δεν θα πρέπει να υπάρχουν γενικές διατυπώσεις γιατί τότε δημιουργούνται προβλήματα. Ενώ αν τα διευκρινίζουμε τότε ε, μεγιστοποιούμε την ασφάλεια για όλες τις επιχειρήσεις χωρίς να παρεμποδίζουμε τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Θελήσαμε λοιπόν λόγω αυτών που συνέβη τον τελευταίο καιρό στον κόσμο, να λάβουμε υπόψη μας περισσότερο και τις φυσικές καταστροφές και θελήσαμε να επιστήσουμε την προσοχή σε ορισμένους τομείς οι οποίοι μας φάνηκαν ότι δεν λαμβάνονταν σωστά υπόψη, μεταφορά επικινδύνων ουσιών και εκμετάλλευση ορισμένων μονάδων είτε πετρελαϊκής παραγωγής είτε άλλων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν φυσικά και σαν ε, χώροι ε, βιομηχανικής δραστηριότητας, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να καλυφθούν και από τη συγκεκριμένη πρόταση. Δεν θα καταθέσω, δεν θα παρουσιάσω όλες τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Θα κλείσω όμως για την μεγάλη ανάγκη που υπάρχει και την οποία εξέφρασαν πολλοί από μας να ληφθούν πραγματικά υπόψη ε, και τα θετικά που προσφέρουν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις. Γιατί φυσικά οι εργαζόμενοι είναι οι πρώτοι που θα αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες, είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα συμμετέχουν άμεσα στις διαδικασίες επεξεργασίας των ουσιών αυτών και θα ήταν σοβαρό πρόβλημα να μην λάβουμε υπόψη μας το ότι θα πρέπει να συμμετέχουν στο σύνολο της διαδικασίας καθορισμού μέτρων ασφαλείας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. Περιμένουμε λοιπόν τώρα και άλλες τροπολογίες και άλλες παρατηρήσεις και είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Η κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ. Εδώ αναπληρώνω τον συνάδελφο Λάζος Μεσάρος που είναι ο σκιώδης ηγητής Δυστυχώ κολλείται σήμερα και μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω και να διαβάσω τα σχόλιά του. Τα προηγούμενα ατυχήματα εξαιτία επικίνδυνων και τοξικών ουσιών μας δίδαξαν ότι αυτός ο τομέας βιομηχανική παραγωγή θα πρέπει να υπόκειται σε έναν αυστηρό μηχανισμό ελέγχου. Και άτυπα δίκτυα μεταξύ επιχειρήσεων και κρατών μελών μπορεί να διαδραματίσουν κέριο ρόλο σε περίπτωση ατυχήματο. Η οδηγία σε Βέζο αυτή τη στιγμή καλύπτει 10.000 μονάδε προκειμένου να αποφευθούν ε, οι κίνδυνοι ατυχήματο. Μία αναθεώρηση θα αυξήσει ελαφρά ε, τον αριθμό αυτών των μονάδων. Τα βασικά στοιχεία της πρότασης είναι τα εξής. Το ίδιο επίπεδο προστασίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται και από την αναθεωρημένη οδηγία με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή είναι η αρχή που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Η παρούσα δεύτερη οδηγία σε Βέζο λειτουργεί καλά. Η αναθεώρηση όμως της οδηγίας αυτής είναι επιθυμητή και για πρακτικούς αλλά και για νομοθετικούς λόγους συνδέεται κυρίως με την ανάγκη ευθυγράμμισης με τον νέο κανονισμό για την ταξινόμηση, σήμαση και συσκευασία των επικίνδυνων ουσιών και σκευασμάτων που θα τεθεί σε ισχύ από το 2015. Μία καλύτερη και ακριβέστερη κατανομή των επικίνδυνων ουσιών και καλύτερη εφαρμογή και προβλεψιμότητα και εκτέλεση των κανόνων είναι προς ε, το κοινό όφελος αλλά και για το καλό του περιβάλλοντος και της βιομηχανίας. Θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των υποχρεώσεων των μονάδων με βάση την συνθήκη και τις επικίνδυνες ουσίες. Επίσης, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι οι διατάξει αναθεωρημένη οδηγία δεν θα πρέπει να υπερβούν το πεδίο εφαρμογή τη. Για παράδειγμα, οι μεταφορέ θα πρέπει να εξακολουθούν να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Αυτή είναι η γνώμη του σκιώδου Σιγητού μας. Οι ρήτρε εξαίρεση των κρατών μελών θα πρέπει να επιτρέπουν κάποια ευελιξία υπό ορισμένε συνθήκε, αλλά θα πρέπει να προβλέπεται ολοσχερή εξαίρεση από την οδηγία. Τα κριτήρια εναρμόνιση για τι εξαιρέσει θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ίδια την οδηγία και να μην ε, προσδιορίζονται σε μεταγενέστερο επίπεδο. Οι πληροφορίες για το κοινό καλύπτονται από την πρόταση. Οι πληροφορίες για μονάδες και κίνδυνο ατυχήματος θα πρέπει να δίνονται στο κοινό και να είναι προσιτές ε, με κατάλληλο τρόπο και στον κατάλληλο βαθμό. Επίσης, ε, τα επίπεδα ελέγχου και πληροφόρησης των κρατών μελών θα πρέπει να εναρμονιστούν για να μειωθεί και το διοικητικό άχθος και κόστος. Ευχαριστώ κυρία Τόγια. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή αλλά και τη γραμματεία που αντιμετώπισαν αυτό το θέμα το οποίο μας οδηγεί στο να κάνουμε κάποιες πολύ ξεκάθαρες βασικές επιλογές προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε και με ποιο τρόπο. Αντιμετωπίζει θέματα επίσης τα οποία πράγματι ε, έχουν ένα επίπεδο τεχνικής δυσκολίας πολύ υψηλό και διαρωτώ με αν μπορούν να συζητηθούν σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα στηρίξουμε τις τροπολογίες του εισηγητή και φυσικά τις δικές μας με τον εξή τρόπο. Όλοι συνειδητοποιούμε ότι και λόγω των τελευταίων συμβάντων που δεν εντάσσονται βέβαια στο πλαίσιο της συγκεκριμένη αυτής πρότασης, αλλά μας εντυπωσίασαν όλους, μας έδειξαν ότι πάρα πολύ συχνά η τεχνολογία και όλα τα συστήματα ασφαλείας ε, είναι τελικά πολύ ευάλωτα και εύθραυστα απέναντι σε κάποια γεγονότα πρόβλεπτα όπως οι φυσικές καταστροφές. Όλα αυτά έχουν αυξήσει το επίπεδο ευαισθησίας μας. Υπάρχει λοιπόν ενδιαφέρον στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα του περιβάλλοντος όπου είμαστε από τις πιο προχωρημένες περιοχές να διατηρήσουμε υψηλό το επίπεδο πρόληψης, αποφυγής και διαχείρισης των καταστάσεων των εκτάκτων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η πρόταση αυτή και για τη δική μας Επιτροπή, όχι μόνο στο επίπεδο του περιβάλλοντος, αλλά θα πρέπει η νομοθεσία να είναι η κατάλληλη κάθε φορά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η αίσθηση ασφαλείας που πρέπει να δώσουμε στον πολίτη θα πρέπει, θα έλεγα, να την χάνουν μια ισόρροπης αντιμετώπισης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συνδυάζοντας όλες τις καταπροτεραιότητες, τις προτεραιότητες τις οποίες έχουμε, την ασφάλεια των εργαζομένων, την ασφάλεια των πολιτών, και μάλιστα χωρίς να αγνοήσουμε και τις θεμητές αν θέλετε απαιτήσει της παραγωγικής πραγματικότητας. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια από πλευράς των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τους εφαρμόσουν σωστά. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα εδώ προτεραιότητας της ασφάλειας, θα πρέπει να την επιδιώξουμε την ασφάλεια και αυτό σημαίνει σαν παράδειγμα ότι κάθε μορφή ενίσχυσης κανόνων οι οποίες καλύπτουν πάρα πολλούς τομείς, οι οποίοι ακόμα και αν δεν καλύπτονται εδώ, είναι κάτι το θετικό. Σαν παράδειγμα και ε, τέτοια στοιχεία στην οδηγία για τις ε, δημόσιες προμήθειες. Και εκεί είναι ένας τομέας ε, στον οποίο θα πρέπει να λειτουργήσουμε με ελεγχόμενο τρόπο, με τρόπο εποπτευόμενο σωστά και δεν θα πρέπει οι κανόνες όταν προκυρήσονται συγγνώμη, διαγωνισμοί για προμήθειες και τα λοιπά να αγνοούνται άλλοι κανόνες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σε ισχύ. Λέγω λοιπόν και προς τον εισηγητή εδώ ότι ε, σχετικά με τις προτάσεις που κάνει για την περιοδικότητα των ελέγχων. Δεν έχει σημασία η συχνότητα και η ποσότητα, αλλά η αυστηρότητα και η εγκυρότητα, η ανάληψη της ε, υποχρέωσης των επιχειρήσεων να σέβονται τους κανόνες και φυσικά η επαλήθευση της, ε, της ε, συγκεκριμένης αυτής υποχρέωσης. Αυτό είναι το καθήκον μας εμάς, όχι να ορίζουμε πολλούς ελέγχους, αλλά να ορίζουμε σωστούς ελέγχους οι οποίοι θα πρέπει να γίνονται με πιο βέβαιο και με πιο αυστηρό τρόπο. Γιατί αν υπάρχουν πάρα πολλοί έλεγχοι, οι έλεγχοι αυτοί είναι ελαφρείς και δεν έχουν βάρος για την σωστή ενημέρωση και αυτό είναι ευαίσθητο θέμα. Η διαφάνεια και η πληροφόρηση είναι κάτι το βασικό. Αλλά όταν υπάρχουν πολλές ενημερώσεις και πολλές πληροφορίες τεχνολογικές, ίσως να μην είμαστε σε θέση να τις χειριστούμε. Κατάλληλη λοιπόν ενημέρωση και στη μορφή και στην ποσότητα. Και εδώ πάλι ανάληψη των ευθυνών από τα αρμόδια όργανα για την επίβλεψη, την εποπτεία και τον έλεγχο της εφαρμογής των κανόνων. Λοιπόν, θα πρέπει να εμείνουμε στο θέμα των ευθυνών, θα πρέπει να υπευθυνοποιήσουμε τα συγκεκριμένα όργανα προστασίας και τότε θα πρέπει να κυκλοφορούν σωστά φυσικά οι ενημερώσεις και οι πληροφορίες. Αν δεν επαρκούν θα τις αυξήσουμε, αλλά δεν πρέπει να προωθούμε συστηματικά την ποσότητα γιατί αυτό θα είναι συχνά εις βάρος της ποιότητας. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει σωστή ενημέρωση και σε εύθετο χρόνο. Αναζητούμε λοιπόν μια ισορροπία. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος, ισορροπία και στον τομέα της ασφάλειας και θα καταθέσουμε τροπολογίες και θα συνεργαστούμε με τον εισηγητή έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταστήσουμε τον χώρο αυτό όσο πιο ασφαλή γίνεται. Ριβάζει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον εισηγητή, τον κύριο Ενά, γιατί έλαβε υπόψη τις συζητήσεις που έγιναν εδώ στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να επιμείνω σε ορισμένα σημεία που αντιμετώπισα και εγώ όταν συμμετείχα σε ένα γενικό έλεγχο στη Γαλλία μετά το ατύχημα του AZF στην Τουλούζη. Το σημαντικό εδώ είναι η ενημέρωση, είπε η συνάδελφος. Να έχετε υπόψη όμως ότι Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ενημερώσουμε τους εργάτες, τους εργαζόμενους. Γιατί αυτή είναι στην πρώτη βαθμίδα της ασφάλειας. Αλλά να ενημερώσουμε και τους ε, γείτονες. Γιατί οι βιομήχανοι δεν ήθελαν να δώσουν τις πληροφορίες ε, στους κατοίκους της περιοχής επικαλούμενοι το εμπορικό απόρριτο. Το θέμα όμως δεν είναι τόσο ποιοτικό όσο ποιοτικό. Φυσικά έχω εμπιστοσύνη στους κατοίκους της περιοχής για να θέσουν τις ερωτήσεις, αλλά και οι βιομηχανοί, οι διαχειριστές θα πρέπει να δίνουν αυτές τις πληροφορίες. Δεν θα πρέπει να περιοριστούμε στο κατέτηση. Όταν έχουμε μία μονάδα σαν το Σεβέζο, θα πρέπει να προβλέψουμε και ένα μηχανισμό και ένα τόπο που θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν τις πληροφορίες, γιατί αν δεν ενημερώνονται, πώς θα ξέρουν ότι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες οι κάτοικοι της περιοχής. Στην Γαλλία έχουμε μια τέτοια υπηρεσία που συνεδριάζει μία φορά το χρόνο και δίνει τις πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους, στον κόσμο που τη ζητάει. Θα πρέπει να προβλέψουμε τέτοιους μηχανισμούς για το πού θα, από πού, από ποια υπηρεσία θα χορηγούνται αυτές οι πληροφορίες. Επίσης υπάρχει και το πρόβλημα της αξιολόγησης των κινδύνων. Στην οδηγία αυτή θα πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση των κινδύνων και από τον αρμόδιο της μονάδας, αλλά υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών και να καθορίσουμε τον περίμετρο της ασφάλειας, γιατί συνήθως έχουμε μια περίμετρο όπου σε περίπτωση ατυχήματος ε, έχουμε κάποιους θανάτους, αλλά θα πρέπει και η περίμετρος της, του ατυχήματος να καλύπτει την περίμετρο της μονάδας και να υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς του γειτονικού οικοπαίδου, γιατί μετά από μία έκρηξη η περίμετρος δεν περιορίζεται στη μονάδα, διευρύνεται πολύ πιο πέρα από αυτήν. Θα πρέπει γι' αυτό να προβλέψουμε αντίστοιχους μηχανισμούς και για τους ελέγχους που είναι πολύ σημαντικοί. Δεν θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε απλώς τους ελέγχους, αλλά να υπάρχει ένα σώμα επιθεωρητών σε κάθε κράτος μέλος αν έχουμε τρει μόνο επιθεωρητέ για τον έλεγχο πολλών μονάδων που εμπίπτουν στην οδηγία τι να το κάνουμε. Θα πρέπει να ελέγξουμε και το σώμα αυτό των επιθεωρητών και να είναι επαρκή. Και μια ανεξάρτητη ε, υπηρεσία για τη βιομηχανία. Πήγα στην Ιαπωνία και είδα πόσε ε, ιαπωνικές αρχές ενδιαφέρονται για την πυρηνική ενέργεια και που υπάγονται στο Υπουργείο Βιομηχανίας. Ξέραμε ότι υπάρχουν κάποιες σύνδεσμοι, και όταν δεν τηρούν, δεν τηρούν οι προδιαγραφές ασφάλειας, υπήρχε δυνατότητα από τις αρχές αυτές να επιβάλλουν κυρώσεις ακόμη και να κλείσουν την επιχείρηση. Θα πρέπει οι αρμόδιες αυτές αρχές να είναι ανεξάρτητες από τους βιομήχανους έχουν, και να έχουν πραγματικές ελεκτικές δραστηριότητες και, και αρμοδιότητες να επιβάλλουν κυρώσεις. Όχι μόνο λόγια να μπορούν οι αρμόδιες αρχές όταν γίνεται η υπέρβαση του κινδύνου και δεν γίνεται σωστή ενημέρωση και υπάρχει κίνδυνος έκρηξης να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους οι αρμόδιες ε, υπηρεσίες γιατί μετά το ατύχημα θα είναι πια αργά θα έχει υποστεί το πλήγμα ο πληθυσμός Σας ευχαριστώ και ας λάβει τον λόγο η Κομισιόν με συγχωρείτε, με συγχωρείτε η κυρία τώρα έχει πάλι τον λόγο. Μία ερώτηση απλή για ένα θέμα το οποίο θεωρώ σημαντικό και για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί πράγματι έχει ήδη δεχθεί κάποιες παρατηρήσεις που εισάγουν καινοτόμα στοιχεία. Είναι το θέμα των εργαζομένων στην επιχείρηση. Νομίζω ότι η πρώτη μας ανησυχία θα πρέπει να είναι για τους εργαζομένους. Δεν υπήρχε αναφορά στους εργαζομένους και το έκανε ο εισηγητής αυτό και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Uh, Σας ευχαριστώ. Ας τα πω στα γαλλικά, μια και οι βουλευτές μίλησαν γαλλικά και ίσως μπορώ να απαντήσω και πληρέστερα. Η Κομισιόν διάβασε με ενδιαφέρον το σχέδιο εκθέσεως του ΣΥΓΙΤΟΥ, παρακολούθησε επίσης με ενδιαφέρον την σημερινή συζήτηση και θα αναφερθώ εδώ σε ορισμένες παρατηρήσεις που συνδέονται και με τις προτάσεις του συγητού και με τη συζήτηση που διεξήχθη. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κοινού, η οδηγία έχει ως στόχο να καθιδρύσει συστήματα πρόληψης αφενός για να διασφαλίζεται ώστε να λαμβάνονται μέτρα πρόληψης στις επιχειρήσεις αλλά ταυτόχρονα να προλαμβάνονται και οι επιπτώσεις των ατυχημάτων. Και εκεί βέβαια τίθεται το θέμα της ενημέρωσης του κοινού. Ε, ε, ενημέρωση που πρέπει να είναι κατανοητή, να μην είναι υπερβαλλόντως τεχνική, να επιτρέψει στους απλούς ανθρώπους να κατανοήσουν τους κινδύνους, καθώς και την στάση που πρέπει να τηρήσουν σε περίπτωση ατυχήματος. Άρα θα υπάρχει τέτοια ενημέρωση για τα ατυχήματα αυτά. Από τη στιγμή που είναι ενήμερο το κοινό, ότι ε, υπάρχει μια επιχείρηση τύπου Σεβέζο να μπορεί να ενημερώνεται και σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο αλλά και σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί. Ο στόχος λοιπόν της ενημέρωσης αυτής θα είναι να είναι ενήμερο το κοινό εφόσον έχει το δικαίωμα αυτό και να ε, γνωρίζει και ποια στάση πρέπει να τηρήσει έχοντας και μια ελάχιστη ενημέρωση για παράδειγμα για τις επιθεωρήσεις που γίνονται οι για τις οποίες μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει τις ε, ευχαριστίες της για την υποστήριξη από τους βουλευτές που μίλησαν σήμερα σχετικά με τις επιθεωρήσεις και είναι γεγονός ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ικανότητα επιθεώρησης ανεξάρτητης στο επίπεδο των χωρών μελών και αυτό είναι πολύ σημαντικό να είναι ανεξάρτητοι οι επιθεωρητές δηλαδή και εδώ αναμένουμε ή μάλλον παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ε, τροπολογίες που κατατίθενται. Η περιοδικότητα των ε, επιθεωρήσεων είναι σημαντική και αυτό στην ε, πρότασή μας δίνουμε τα ελάχιστα κριτήρια ανατολισμούς των επιθεωρήσεων για εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου μία φορά τον χρόνο και για χαμηλότερο κινδύνου μία φορά ανά τριετία. Για μας τα μέτρα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά για να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της οδηγίας. Διότι όσοι όλοι γνωρίζουν, το επίπεδο ασφαλείας που επιτυγχάνεται σε μια εγκατάσταση μπορεί σιγά σιγά να αποδυναμωθεί, μπορεί να επιδεινωθεί, διότι τα μέτρα ίσως δεν τηρούνται απολύτως. Χρειάζεται λοιπόν ε, τακτικές επιθεωρήσεις και επισκέψεις επιτόπου ενδεχομένως με την συμμετοχή και των εργαζομένων. Και αυτό με φέρνει στο θέμα που ετέθη σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων. Βέβαια, υπάρχει η οδηγία πλαίσιο που εφαρμόζεται στις δραστηριότητες αυτές, όπως το διαλαμβάνουμε και στο προήμιό μας, είναι η 89391 η οποία διαλαμβάνει διάφορα μέτρα για τις ε, ενώσεις εργαζομένων και θα δούμε τις τροπολογίες βέβαια και σε ό,τι αφορά την προστιθέμενη αξία. Για μας είναι και εκτιμένο ότι οι, οι εργαζόμενοι πρέπει να παίξουν ένα ρόλο. Να δούμε όμως ποιος θα είναι, ποια θα είναι μάλλον η προστιθέμενη αξία της συμμετοχής αυτής. Γιατί καμιά φορά υπάρχουν αποκλήσεις μεταξύ των νομοθετικών μέτρων Πάντω επί τη ουσία δεν, δεν έχουμε πρόβλημα με την νομοθεσία αυτή. Και ε, εξ για δύο ή τρία σημεία όπου έχουμε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της έκθεσης για την αποζημίωση των θυμάτων. Πρώτα, που απορρέει από την ε, από το αστικό δίκαιο που εφαρμόζεται στις χώρες μέλη. Εκεί δεν μπορούμε να παρέμβουμε και δεν θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να, να ληφθούν μέτρα για θέματα αποζημίωσης που όπως είπα τα προβλέπουν τα δίκαια των χωρών μελών που είναι άλλωστε και οι κατάλληλες οι χώρες μέλη δηλαδή για να ρυθμίσουν τα σχετικά. Υπάρχει και μια τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα για τις προθεσμίες μέσα στις οποίες ορισμένες εγκαταστάσεις οι οποίες θα ε, εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να συμμορφώνονται. Βεβαίως ένας επιχειρηματίας μπορεί να αποφασίσει να κάνει κάποιες αλλαγές στις εγκαταστάσεις του και να, και να εμπέσει σε κατηγορία τύπου σεβέζου. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί χρόνος για να γίνει αυτό και νομίζω ότι στο τεχνικό επίπεδο χρειάζεται κάποιες διευκρινήσεις σε συνεργασία με τον εισηγητή. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας υπάρχουν ορισμένες προτάσεις που γίνονται διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογή. Πρώτα τίθεται το θέμα του στρατιωτικού τομέα. Γνωρίζετε ότι η συνθήκη προβλέπει ιδιαίτερε ε, διατάξεις για τα στρατιωτικά για τον κίνδυνο ατυχήματος που αυτά βέβαια τα διαχειρίζεται το ίδιο το ε, στατιωτικό ε, πλαίσιο για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και δεν μπορεί να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή οδηγία μα. Αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί έτσι. Σε ό,τι αφορά τι μεταφορέ. Αναγνωρίζουμε ότι οι μεταφορέ είναι σημαντικό θέμα. Μεταφορά δηλαδή επικινδύνων ουσιών που προκαλούν κινδύνους και που δεν είναι του ίδιου τύπου οι κίνδυνοι αυτοί όπως με μια σταθερή εγκατάσταση. Ε, έχουμε δει βέβαια τα τελευταία χρόνια και ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζεται μέχρι τώρα θεωρούμε ότι είναι ο καταλληλότερος. Κύριε Πρόεδρε, 30 δευτερόλεπτα ακόμη για να έλθω στο θέμα των αγωγών, pipelines, καθώς και τις ε, υπεράκτης εγκαταστάσεις, offshore, για τους αγωγούς, η Κομισιόν διεξάγει μελέτη σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από την χρήση αυτών των εγκαταστάσεων. Θα χρειαστούν λίγοι μήνες ακόμη μέχρι ότου ολοκληρωθεί η μελέτη αυτή και στη βάση των πορισμάτων της μελέτης αυτής θα ε, βγάλει συμπεράσματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή για τις εγκαταστάσεις εξόριξης πετρελαίου, offshore. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εξέδωσε ανακοίνωση πέρσι και για φέτος προτιθέμεθα να ρυθμίσουμε συγκεκριμένα τα περιβαλλοντικά μέτρα για τις ε, ε, δεξαμενές αυτές. Χρειάζεται ένας μηχανισμός πιο ειδικό για τις δραστηριότητε αυτές που ε, παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Ο κύριος Όντι. Σύντομα, Πρόεδρε, θα συγχαρώ τον εισηγητή και να επιστήσω την προσοχή του σε κάτι το οποίο ίσως να καλύπτεται βέβαια από συγκεκριμένα άλλα εγγραφά ότι οι επιχειρήσεις αυτές, οι εγκαταστάσεις αυτές είναι σωστά ασφαλισμένες όταν αυτό το μείζον τύχημα το οποίο προβλέπεται από όλες αυτές τις προφυλάξεις συμβεί. Αν δούμε σαν παράδειγμα την καταστροφή της εξέδρας της British Petroleum θα δούμε ότι είναι μία από τις λίγες εταιρείες που ασφάλιζε μόνη της την εγκατάσταση. Βέβαια ήδη οι πόροι της επιχείρησης και οι αποζημιώσεις βέβαια δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά ήδη οι πόροι της επιχείρησης καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις θα ήθελα να υπάρχει ένα συγκεκριμένος έλεγχος, έτσι ότι είτε με ιδίους πόρους, είτε με συγκεκριμένα ασφαλιστικά συμβόλαια, με ε, θα έλεγα ικανές να καλύψουν το κόστος ασφαλιστικές εταιρείες, να υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των ζημιών αυτών, έτσι ώστε αυτές οι ζημίες που μπορεί να είναι μεγάλου μεγέθους να μην επηρεάζουν τα δημοσιονομικά γιατί τελικά το συνολικό κόστος της εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων αυτών πρέπει να περιλαμβάνει και όλες τις συνέπειες σε επίπεδο ασφαλείας. Ο κύριος Σενά, θέλετε εκ νέου το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βλέπουμε ότι τα πράγματα προχωρούν. Ο ρόλος μας όπως βουλευτές είναι να πιέσουμε έτσι ώστε να έχουμε περισσότερη ασφάλεια στις κοινωνίες μας είναι λοιπόν καθήκον μας να κάνουμε προτάσεις οι οποίες και δεν θα ληφθούν ίσως αμέσως υπόψη, βοηθούν το σύστημα να προδεύσει και να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών. Μιλάμε για την ασφάλεια των ανδρών και γυναικών που εργάζονται στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, ε, των κατοίκων της περιοχής, τη συγκεκριμένη αν θέλετε επιχείρησης, γιατί όταν χάνεται ένα μέσο παραγωγής χάνεται και ο πλούτος που το δημιούργησε. Είναι απαραίτητο λοιπόν να καλύψουμε όλους τους τομείς ασφαλείας, όπως είναι απαραίτητο και να μιλήσουμε και για τους ελέγχους, αλλά κυρίως για την αυστηρή τους εφαρμογή. Γιατί αν πράγματι γίνεται ένας έλεγχος και δεν υπάρχουν κυρώσεις σε αυτούς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσει, τότε δεν θα προχωρήσουμε. Είναι λοιπόν απαραίτητο πρώτο να επιτρέψουμε στην διαδικασία τη βιομηχανική να συνεχιστεί, αλλά να δώσουμε τη δυνατότητα και στους κακούς μαθητές να επανέλθουν στην τάξη και να ανταποκριθούν στους κανόνες. Κατά τα άλλα θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και περιμένω τις τροπολογίες με πολύ πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ κύριε Ένα. Προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών η 6η Εβδόμου. Μα το είπα. Μόλις τώρα. 6 Ιουλίου για τις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ όλες και όλους. Λίγη εδώ το θέμα υπαριθμών 8 της ημερησίας διατάξεως. Υπάρχουν τα διάφορα. Δεν έχω τίποτε στα διάφορα και τόσο το καλύτερο. Το 10 τα διαβάζετε πότε θα γίνουν οι επόμενες συνεδριάσεις. Εδώ λοιπόν λίγη η συνεδρίαση.